Αγαπητοί φίλοι, ας ξεκινήσουμε για εργασία της Επιτροπής. Bene. In considerazione della riunione straordinaria. Όσον αφορά την έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Γεωργίας που προβλέπεται να διεξαχθεί στις 5 Οκτωβρίου ή την επόμενη Δευτέρα, θεώρησα χρήσιμο να προσθέσω στη σημερινή μερίσια διάταξη το θέμα της κρίσεως του γαλακτοκομικού τομέα όπως τα κράτη-μέλη ζήτησαν να συζητηθεί η δυνατότητα να παρέμβουμε για υποστήριξη του τομέα και με άλλα μέτρα. Και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει πλήρως στην διεξαγωγή της συζήτησης. Κυρίως μετά από την υιοθέτηση του ψηφίσματός μας που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα εις Στρασβούργων, σήμερα μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις επί του θέματος και να ακούσουμε τι συνέχεια προτίθεται να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ψήφισμά μας. Λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τις προτάσεις ε, που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη. Ρωτώ αν συμφωνείτε να το βάλουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και ρωτώ αν είναι δυνατόν να μεταθέσουμε το σημείο για την ποιότητα, την ποιοτική πολιτική του κυρίου Σκότα που θα κάνει την ανακοίνωση θέλει, αν είναι δυνατόν, να το εξετάσει το θέμα αυτό στο τέλος της μερίσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, η μερίσια διάταξη εγκρίνεται με τις προταθήσεις αλλαγές. Καλώς. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω σε τι αναφερόσατε. Σήμερα, σήμερα λέτε ότι θέλετε να το εξετάσουμε. Σήμερα το απόγευμα. Εντάξει. Μάλιστα, μάλιστα. Στο τέλο μόνο, για να επιτρέψω τον κύριο Σκότα ε, που θα έρθει αργότερα να μπορέσει να μα ενημερώσει ε, με περισσότερε λεπτομέρειε. Έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, πριν το τέλο τη σημερινή συνεδριάσεω, τα πρακτικά θα θεωρηθούν ω εγκεκριμένα. Σας ενημερώνω ότι η σημερινή συνεδρίαση μεταδίδεται και στην αίθουσα ακρόασης στην ASP 5G3. Καλώς. Η κατάσταση του γαλακτοκομικού τομέα και τα δεχόμενα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν βραχυπρόθεσμα και μέσο πρόθεσμα. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής Θέλαμε μέσω της κυρίας Φίσερ της Επιτρόπου, στις 17 του μηνός που πέρασε, συζητήσαμε το θέμα και εκτιμήσαμε την προσοχή που προσδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο, που ήρθε και μας παρουσίασε η Επίτροπος ε, νέες πρωτοβουλίες, νέες προτάσεις για το γαλακτοκομικό τομέα. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Σμούσεν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας ενημερώσει λεπτομερέστερα όσον αφορά το περιεχόμενο των νέων προτάσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλό θα ήταν να σα ενημερώσω όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τονίσω επίσης τη σημασία που έχουν αυτές οι πρωτοβουλίε και από τη συμφωνία που ενεκρίθη με μεγάλη πλειοψηφία και από το ψήφισμα. Και με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε και η πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, η δική μας, που εγκρίθηκε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας ομόφωνα. Υπογραμμίσαμε σε αυτή την περίσταση και στην παρέμβασή μου και ευχαριστώ όσους μίλησαν επίσης στην Ολομέλεια του Στασβούργου, λέγω, υπογράμμισα ότι το θέμα είναι ένα θέμα όχι μόνο θέμα μηνύματος που θα απευθύνουμε προς τους γαλακτοπαραγωγούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και θέμα πολιτικής φύσεως. Δεν θα σας διαφεύγει ότι αν την επόμενη εβδομάδα το δημοψήφισμα η Ιρλανδία είναι θετικό, όπως όλοι ευχόμεθα, θα εισέλθουμε στην εποχή της συναποφάσεως. Είναι προφανές λοιπόν ότι το πρώτο Συμβούλιο Υπουργών που θα λάβει η χώρα της Λουξεμβούργο 19 και 20 επόμενου μήνος και που θα λάβει αποφάσεις για το γαλακτοκομικό και τυροκομικό τομέα θα πρέπει να εξετάσει με μέγιστη προσοχή της, ε, τη δική μας νομοθετική πρόταση. Και γι' αυτό σήμερα το πρωί μαζί με τους συντονιστές όλων των ομάδων της Επιτροπής μας δεχθήκαμε το αίτημα του Γάλλου Υπουργού, του κυρίου Λεμέρ, να έρθει και να μιλήσει όσον αφορά την γάλλο-γερμανική πρωτοβουλία που ακολούθηκε για άλλους 18 υπουργούς. Σήμερα το έγγραφο υπογράφεται από 20 υπουργούς. Και μας παρουσίασε ο υπουργός τις ιδέες που αυτή η ομάδα τουλάχιστον των 20 υπουργών, τις ιδέες που θα προτείνουν αυτοί οι υπουργοί στο επίσημο ε, συμβούλιο που θα γίνει 19 ε, και 20 Οκτωβρίου. Με χαρά μου λοιπόν δίνω το λόγο στην κυρία Ρασμούσεν και μετά καλό να ακουστούν και κάποιες σκέψεις. Δεν θα ασχοληθούμε όλο το απόγευμα βέβαια, αλλά θα ήταν χρήσιμο να υπογραμμιστεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου, ο δικός μας ρόλος σε αυτή την ευαίσθητη και δύσκολη κατάσταση που περνά ο γαλακτοκομικός ε, τομέας. Ρασμούσεν. Ο κύριος Δασμούσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά στοιχεία του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου του Στρασβούργου ήταν να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο τακτικά να παρέχει πληροφορίες όσον αφορά την αγορά και όσον αφορά τον γαλακτοκομικό τομέα. Ξεκινώ από εκεί, από τα θετικά στοιχεία, όπως υποσχεθήκαμε στο Συμβούλιο Γεωργίας, να δίνουμε κάθε τρεις μήνες ε, αναφορά για την κατάσταση αγοράς, μπορούμε να δεσμευτούμε εξίσου να διανέμουμε αυτή την έκθεση για την αγορά και στα μέλη της Επιτροπής σας. Δεν είναι έτοιμη η έκθεση. 19 Οκτωβρίου θα είναι έτοιμη η έκθεση για το Συμβούλιο. Αλλά θα ήθελα σήμερα ε, να σας δώσω κάποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση αγοράς σήμερα από το μήνα Ιούνιο. Είδαμε μία ανάκαμψη των τιμών, έχουμε καλύτερες τιμές. Αυτό Το ότι βλέπουμε στην παγκόσμια αγορά καλύτερε τιμέ στην παγκόσμια αγορά καθώ και στην εσωτερική αγορά είναι κάτι ενθαρρυντικό. Και ελπίζουμε ότι δεν είναι κάτι παροδικό και δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά είναι η αρχή μιας καλύτερης ε, τάσης για τον γαλακτοκομικό τομέα. Να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Οι τιμές του γάλακτος στην Ολλανδία αυξήθηκαν κατά 50% από το μήνα Ιούνιο. Spot in Στη Βόρεια Ιρλανδία 19 με 20. Το προηγούμενο ποσοστό μάλλον ήταν 15 διορθώνει Ιταλία περίπου 12%. Βλέπουμε ποιε είναι οι τιμές αγορά. Είναι τιμέ ανοιχτέ τιμές είναι τιμές spot. Πρέπει να, και, να δούμε και τι γίνεται με τη ζήτηση σήμερα. Είναι μεγαλύτερη η ζήτηση τώρα, σχετικά, μεγαλύτερη ζήτηση γάλακτος τώρα από την προμήθεια. Τώρα όσον αφορά τις τιμές του γάλακτος, επισυμβατικής βάσεως, αυξάνονται σε όλες τις μεγάλες παραγωγές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η πρώτη ύλη, το γάλα, η τιμή του γάλακτος αυξάνεται. Ακούμε αυξήσεις 1 με 2 cents το λίτρο, από 25 cents πήγαμε στα 27 cents το λίτρο. Σε μια μεγάλη χώρα όπως η Γαλλία, όπως και 28 cents ανά λίτρο. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι ενθαρρυντικό. Απέχει πολύ από την τιμή παρέμβασης που είχαμε πολύ παλιά, 21,5 και καλύτερα από το 23 και 24 κατά μέσο όρο που είχαμε τιμή τον Ιούνιο. Παρενέβημεν και για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την αγορά στο βαθμό του μέτρου και να βοηθήσουμε την αύξηση των τιμών και θέλουμε να υποστηρίξουμε έχουμε βγει την παρέμβαση να αφορά το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη οι τιμές παρέμβασης του βουτύρου είναι 2.218, η τωρινή τιμή είναι 2.380 για το βούτυρο. Περίπου κοντά στην τιμή παρέμβασης. Αυτή είναι η, κατάλη, η κατάσταση τελευταία, τελευταίους δύο μήνες. Το ίδιο για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Είδαμε μια αύξηση στους τρεις μήνες του 9%. Πάνω από την τιμή παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη περίπου κατά 6%. Το γάλα σε σκόνη ε, έχει αυξηθεί κατά 9% και το τσένταρ, το τυρί τσένταρ, έχει αυξηθεί κατά 5%. 5%. Αυτά είναι τα θετικά μηνύματα της ε, αγοράς, της κοινοτικής αγοράς. Στην παγκόσμια αγορά τώρα, που και αυτό είναι σημαντικό, και πρέπει οι εξαγωγείς μας να μπορούν να πουλήσουν στην παγκόσμια αγορά και να έχουν καλά κέρδη από την παγκόσμια αγορά και είναι και θέμα ψυχολογικό ότι πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ψηλές τιμές στην παγκόσμια αγορά. Μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά το βούτυρο, σε σχέση με τις αναφορές από Λιθουανία και από, Νέα, από Ζηλανδία μάλλον, που βασικός εξαγωγέας, βλέπουμε ότι αυξήθηκαν τιμές του βουτύρου κατά 19% από τον Ιούνιο. Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη 10% γάλα σε σκόνη, πλήρες γάλα, κατά 24%. Αλλά για κάποιο πλήρες γάλα σε σκόνη που πουλείται σε δημοπρασία, μηνιαία, αυτές οι τιμές αυξήθηκαν κατά 51% και τιμές για αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη στις ΙΠΑ και εκεί είδαμε πριν από 6-12 μήνες ΙΠΑ ήταν μεγάλος ανταγωνιστής λόγω χαμηλών τιμών και μεγάλου διαθέσιμου όγκου στην παγκόσμια αγορά. Δεν ισχύει πια αυτό. Οι τιμέ για αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη αυξήθηκαν και ο όγκο προ εξαγωγή από τη ΣΥΠΑ μειώνεται δραματικά. Νομίζω λοιπόν, Πρόεδρε, ότι αυτά είναι κάποια στοιχεία που σας παραθέτω για να σας δείξω πού βρισκόμαστε σήμερα, αλλά ίσως πιο σημαντικό, ποια τάση ε, δημιουργείται και σε ποια τάση κινούμαστε, ακολουθούμε σήμερα. Αναφερθήκατε στην παρέμβαση της Επιτρόπου μου στην, ε, στο Στρασβούργο και αναφερθήκατε και στο ψήφισμα των 30 σημείων που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορώ σήμερα, διότι δεν έχω εντολή, δεν μπορώ λέω σήμερα να επισέλθω σε λεπτομέρειες σχετικά με κάθε σύσταση που συμπεριλάβατε στο ψήφισμά σας. Όμως είναι εξίσου σαφές ότι διαβαστούν μετά της δέουσας προσοχής και θα εξεταστούν δεόντως. Κάποια από αυτά τα σημεία, Πρόεδρε, ε, ταιριάζουν, είναι παράλληλα με τις συστάσεις της ομάδας των 20. Η δήλωση που ήταν πρωτοβουλία γαλλογερμανική και υπεγράφει από άλλους 18 κράτη-μέλη, από άλλα 18 κράτη-μέλη, αυτές οι συστάσεις θα συζητηθούν, θα αξιολογηθούν προσεκτικότατα και φαντάζομαι ότι η πρώτη ευκαιρία να γίνει κάτι τέτοιο θα είναι στο άτυπο Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου, την επόμενη Δευτέρα, όπου η Επιτροπός μου θα συναντήσει τους συναδέλφους από τα 27 κράτη-μέλη σε ένα ανεπίσημο γεύμα. Το γεύμα δεν θα κρατήσει πάνω από ένα δύο ώρο, ήθιστε αυτό για ένα γεύμα, κανονικό διάστημα. Και φαντάζομαι επίσης ότι οι Υπουργοί και οι Επίτροπος δεν θα μπορέσουν να επισέλθουν σε πολλές λεπτομέρειες. Όμως θα μπορούσαν να καταλήξουν σε προσανατολισμούς για το πρακτέον. Και όπως είπε η ίδια Επίτροπος στο Στασβούργο, προτίθεται να ζητήσει υποστήριξη για την συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου για να εξετάσουν αυτά τα θέματα. Μέσω μακροπρόθεσμα, από μία μέσω μακροπρόθεσμη σκοπιά. Και υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα προς συζήτηση. Αυτά για το άτυπο συμβούλιο. Η, η Επίτροπος και το άτυπο συμβούλιο θα καταλήξουν σε προσανατολισμούς και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προσανατολισμών, γνωρίζοντας ότι εξακολουθεί η κρίση, παρά τα όσα παρέθεσα όσον αφορά τις θετικές τάσεις, εξακολουθεί να υφίσταται κρίση, η, ο γαλακτοκομικός τομέας, η γαλακτοπαραγωγή ε, δεν είναι ικανοποιητική, δεν είναι ικανοποιημένη, συγγνώμη. Άρα κάτι πρέπει να γίνει. Υπήρξε συμφωνία με την πρόταση παράταση παρέμβαση για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Θέλουμε να παραμείνει ανοιχτό το πεδίο. Παρά το γεγονό ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή παρέμβαση, αλλά θα το κρατήσουμε αυτό σαν ένα μέσο, ένα εργαλείο, ενεργό εργαλείο, αν χρειαστεί. Αν οι τάσεις αντιστραφούν και κινηθούμε ξανά προς τα επίπεδα παρέμβασης. Επαγρυπνούμε. Χρησιμοποιούμε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις ε, όσο πιο πολύ μπορούμε, τις εξαγωγικές επιστροφές μάλλον. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί ε, λόγω συμφωνιών με τον ΠΟΕ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε ή ό,τι θα θέλαμε να κάνουμε ή ό,τι θα ήθελε να κάνουμε ο γαλακτοκομικό τομέα. Υπάρχουν διεθνεί περιορισμοί και πρέπει να συμμορφωθούμε και με αυτού του περιορισμού και τα ωρία. Επ' αυτή τη βάση, λοιπόν, τα βραχυπρόθασμα μέτρα τα μέτρα καθημερινής στήριξης εξακολουθούν να υπάρχουν, χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται από τους εμπλεκομένους φορείς, από αυτούς που κατεργάζονται τα προϊόντα και τους εξαγωγείς για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Τι θα εξετάσουμε λοιπόν. Μέσω μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Όσον αφορά κάποια από τα σημεία που συμπεριλάβατε στο ψήφισμά σας και κάποια σημεία που έχουν θίξει και οι υπουργοί στην κοινή τους δήλωση. Πρόεδρε, νομίζω ότι δεν θα πω περισσότερα σε αυτό το στάδιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίες της είναι πολύ ανοιχτή, επιδεικνύει ανοιχτό ανοιχτό πνεύμα όσον αφορά τα όσα προτείνονται. Είμαστε συνεργάσιμοι και βλέπουμε αποτελέσματα. Για να τα βάλουμε όλα στο σωστό πλαίσιο. Βλέποντας την αύξηση των τιμών. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι τιμές spot. Αυτές που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση μακροπρόθεσμες συμβάσεις, αυτές οι τιμές δεν είναι γνωστές σε εμάς. Και ίσως εδώ έγκυται το πρόβλημα. Ότι οι μεταποιητές του γάλακτος χρησιμοποιούν γαλακτοκομικά προϊόντα που κατά 75-80% από το γάλα που παράγεται πωλείται στο λιανεμπόριο με τον ένα τον άλλο τρόπο. και η τιμή στη λιανική μπορεί να μετατραπεί σε υψηλότερη τιμή γάλακτο αμέσω ή με χρονική στέρηση διμήνου τριμήνου. Αυτό εξαρτάται από τι διαπραγματεύσει Τη διάρκεια τη σύμβαση μεταξύ των δύο μερών είδαμε κατά το παρελθόν το 2007 όταν άρχισαν να αυξάνονται οι τιμε χρειαστηκαν Χρειάστηκαν τρει-τέσσερι μήνε μέχρι ότου να ακολουθήσουν και οι, να ακολουθήσουν οι μέσες τιμές, ο μέσος όρος. Εδώ αυξάνονται οι τιμές των γαλακτοκομικών, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει χρονική υστέρηση. Ότι ο χρόνος για να αυξηθεί ο μέσος όρος της τιμής δεν χρειάζεται τρει-τέσσερι μήνες πλέον, αλλά μικρότερο χρονικό διάστημα. Πρέπει να καταλάβουμε αυτή την αντίληψη, αυτό, αυτή την εικόνα σχηματίζουμε από πλευράς του λιανεμπόριου. Και αυτοί το ίδιο πιστεύουν. αυτά που είπα ισχύουν και για τους ε, μεταποιητές και για τους ε, παραγωγούς, τους γαλακτοπαραγωγούς. Καλώς. Ευχαριστούμε. Τον κύριο Ρασμούσεν. Θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε λεπτομερέστερα ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα υποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Να ξεκαθαρίσω προ τον κύριο Ρασμούσεν αλλά σε όλου μα ότι υπάρχει ένα ψήφισμα που με μεγάλη πλειοψηφία θετήσαμε. Και υπάρχει και μια πρόταση νομοθετική συγκεκριμένη που ενέκρινε αυτή η Επιτροπή που δεν έχει την ίδια αξία. Θα ανοίξουμε τη συζήτηση. Ήδη έχω εγγράψει 12 μέλη που θέλουν το λόγο. 13 τελευταία, τελευταίος που εγγράφεται χειριστείτε σωστά τον χρόνο. Μας έφαγαν χρόνο και συντονιστέ που τους άφησα πολύ χρόνο. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Για την ώρα δεν καθορίζουμε κάποια συγκεκριμένη διάρκεια, αλλά πώ να το πω, βασίζομαι στην καλοσύνη. Albert Des. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι φαίνεται να μειώνεται κάπως η ένταση στις αγορές. Μίλησα πριν με τον πρόεδρο των ενώσεων γαλακτοπαραγωγών στην ε, πατρίδα μου και επιβεβαιώνει αυτά που είπε και ο κύριος Ράσμουσεν ότι υπάρχει μια ανωδική τάση των τιμών. Ωστόσο, επισημαίνω και σε εσά κύριε Ράσμουσεν αυτό που είπε και ο πρόεδρος μας ότι ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο ψήφισμα με μεγάλη πλειοψηφία και καλώς θα πράξει η Κομισιόν να λάβει σοβαρά υπόψη τα σημεία που περιλαμβάνει το ψήφισμα αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα συμμετέσχα σε συνάντηση με την Επίτροπο κυρία Φίσερ Μπόουλ και έμαθα εκεί, αν και το γνωρίζαμε ήδη από πριν, ότι πρόκειται να κατατεθεί πρόγραμμα για να χρησιμοποιηθούν γαλακτοκομικά προϊόντα και στην ε, και περισσότερα στην ε, βιομηχανία παραγωγής παγωτών ε, και σε άλλες. Στην αγροτική πολιτική υπάρχουν μηχανισμοί που δεν θα πρέπει να καταργηθούν αυτομάτως. Ας μπουν σε μηδενική βάση ώστε να τους έχουμε στη διάθεσή μας εφόσον χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κρίσεως. Ήταν βαρύ σφάλμα που καταργήθηκαν κάποιοι μηχανισμοί. Πρέπει να διατηρούνται οι μηχανισμοί, διότι εάν καταργηθούν και χρειαστούν μετά σε μια κρίση, πρέπει να ξαναψηφιστούν και είναι απαραίτητο να βρεθούν οι πλειοψηφίες. Ίσως αυτό είναι ένα θέμα πιο πολύ εθνικό. Αλλά, όπως και να έχει το πράγμα, πρέπει οπωσδήποτε να μπορούμε να χρηματοδοτούμε εθνικά μέτρα επίσης. Συγχρηματοδότηση να υπάρχει για αυτά τα μέτρα. Έγιναν συνεδριάσεις στη δικιά μου εκλογική περιφέρεια, όπου πολλοί παραγωγοί κάπως πιο μεγάλοι στην ηλικία, ήρθαν και μας ρώτησαν αν πάλι υπάρχει αυτός ο κανονισμός ε, που απευθύνεται στους αγρότες ε, μεγαλύτερης ηλικίας από τα 55 και σκέφτονται να πάρουν πρόορη σύνταξη. Χρειάζονται εκεί για τους ανθρώπους αυτούς να προβλεφθούν ειδικά προγράμματα με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως εφόσον, εφόσον γίνει αυτό θα ε, μειωθεί η ένταση και η κατάσταση τώρα για την ε, αγορά. Εγώ είμαι στο Προεδρείο μιας μεγάλης ομοσπονδίας γαλακτοπαραγωγών. Τους τελευταίους μήνες αναγκαστήκαμε διότι έχουμε και να μετακινήσουμε τις ποσότητες αυτές χρειάστηκε να κάνουμε συμβάσεις σε αιτήσια βάση και μας απείλησαν ότι θα μας διαγράψουν από τις λίστες τους ορισμένοι, ορισμένες, ε, ε, ορισμένοι αντισυμβαλόμενοι που είπαν ότι θα μας διαγράψουν από τις λίστες τους εάν δεν κάνουμε ε, συμβάσεις σε αιτήσια βάση μαζί τους. Ένα μεγάλο μέρος λοιπόν της παραγωγής χρειάστηκε να περάσει έτσι. Το 2007 όπου ήταν υψηλές οι τιμές και όπου εμείς θα θέλαμε βέβαια τότε να υπάρξουν συμβάσεις σε βάση ετήσια τότε ε, οι μεγάλοι αυτοί καταναλωτές γάλακτος μας είπαν όχι μέχρι τρεις μήνες για να μπορούν να υποφεληθούν από μια ενδεχόμενη κατόπιν μείωση της τιμής. Πάντω αυτά που μας περιμένουν είναι σημαντικέ προκλήσεις για όλους μας και πρέπει να δώσουμε σοβαρή προσοχή. Καπούλα έχει Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και αρκετού μήνε, Πρόεδρε, επικρίνω την Εκτελεστική Επιτροπή. Και γιατί. Επειδή έχει μια κατάσταση δημιουργήσει που πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από τα μηνύματα που παίρνουμε από την αγορά. Το να δίνουμε την εντύπωση στην αγορά ότι μπορεί να αυξάνει την παραγωγή χωρίς όρια ήταν σφάλμα. Οι τιμές είχαν ήδη αρχίσει να μειώνονται, ενώ η Επιτροπή κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένει η αγορά από μόνη της να λύσει το πρόβλημα. Συγχρόνως δε, πολλές ε, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αναγκάζονται να κλείσουν. Αυτή η κρίση, εγώ είμαι πεπισμένος ότι είναι συγκυριακή κρίση. Και ακριβώς είναι συγκυριακή και ακριβώς επειδή είναι συγκυριακή και προσωρινή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε αμέσως και όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάρει μέτρα για να υπάρξει αύξηση. Διότι βλέπετε το γάλα δεν είναι όπως τα αυτοκίνητα όπου μπορούμε να στείλουμε δύο μήνες τους εργάτες στο σπίτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει πάει πιο μακριά, θα έπρεπε να έχει κάνει περισσότερα με επιπλέον ενισχύσεις ώστε η παραγωγή να μπορούν να παράγουν λιγότερο. Εγώ περίμενα από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής κάτι παραπάνω μπορεί να μην έφερνε καινοτομίε, αλλά αν μη τι άλλο τον ε, Οκτώβριο να έρθει να μας πει κάτι παραπάνω πριν από την συνεδρίαση των Υπουργών στις 20 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο, ανάμεσα στις 5 και τις 20 Οκτωβρίου δηλαδή, να έρθει να μας πει τι μέτρα σκοπεύει να προτείνει η Επίτροπο στο Συμβούλιο. Και για να δούμε επίσης μήπως τελικά καταλάβουμε τι θέλει να κάνει η Επίτροπος. Θα κάνει κάτι σοβαρό ή απλώς θα κερδίσει χρόνο με το τίποτα. Σας ευχαριστώ Λουίς. Αντιπρόεδρος Νικολέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτα απ' όλα, μία γενική παρατήρηση και μία πιο συγκεκριμένη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί το θέμα του γάλακτος έχει βρεθεί στα πρωτοσέλιδα τον τελευταίο καιρό. Είναι αλήθεια ότι η κρίση είχαμε σε ολόκληρη τη γεωργία και σε ολόκληρη σε όλους τους οικονομικούς ε, τομείς. Στη δικιά μου τη χώρα, τη Ρουμανία, φέτος οι αγρότες είχαν 5 εκατομμύρια ε, συγκομιδή ε, δημητριακά 400 με 500 ευρώ ανά εκτάριο και ο μέσος όρος ήταν 70 με 90 ευρώ. Οι αγρότες λοιπόν στη Ρουμανία κατέγραψαν μία μείωση 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Οπότε η κρίση δεν ε, πλήττει μόνο τον γαλακτοκομικό τομέα και εμείς με το σιτάρι έχουμε τεράστιο πρόβλημα στη Ρουμανία που αξίζει τον κόπο να το κοιτάξουμε. Και είναι εξίσου σοβαρό το πρόβλημα όπως και εκείνο με το γάλα. Τώρα μια πιο συγκεκριμένη παρατήρηση που έχω να κάνω. Τον τελευταίο καιρό Μίλησα για τα μέτρα ενθάρρυνσης της γαλακτοκομικής παραγωγής. Στο ψήφισμα που εγκρίναμε στο Στρασβούργο αναφέραμε μια λύση. Όμως δεν αναρωτιόμαστε περιορίστε στο χρόνο η λύση αυτή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υποφελούνται από τη ρύθμιση αυτή όχι μόνο οι γαλακτοπαραγωγή αυτή, αλλά και αυτοί που μεταποιούν το γάλα στη συνέχεια. δεν ενθαρρύνουμε τη ζήτηση αν και ο παραγωγός δεν έχει αύξηση στις τιμές. Πιστεύω λοιπόν ότι το γάλα που πηγαίνει στα σχολεία, γιατί αυτή ήταν η λύση που είχαμε προτείνει, πρέπει να παράγεται με σωστό τρόπο. Στη Ρουμανία ένα ποτήρι γάλα στα σχολεία έχει μεγαλύτερη τιμή από όσο πληρώνουν οι γονείς για ένα ή για δύο λίτρα γάλα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μια τέτοια λύση είναι υπέρ των παραγωγών. Πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε αυτό το σύστημα, να σκεφτούμε το σωστό, το δίκαιο εμπόριο. Αλλιώς καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αυτή με τα σχολεία και το γάλα που δίνουμε στα σχολεία είναι ένα σύστημα από το οποίο υποφελούνται οι μεταπητές και όχι οι ίδιοι παραγωγοί γάλακτος. Ευχαριστώ και Νικολέσκου. James Nicholson, επόμενος θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όλοι πρέπει να καλωσορίσουμε την πρωτοβουλία σα για τη διεξαγωγή τη συζήτηση σήμερα το απόγευμα μετά τη συνάντησή μα που είχαμε το Γάλλο Υπουργό σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο το να συζητήσουμε τα θέματα τώρα. Σίγουρα σημείωσα ότι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε επιστροφή σε καλύτερε τιμέ, όπω είπε και η Επίτροπο την περασμένη εβδομάδα. Ακόμα και για τη Βόρεια Ιρλανδία, την περιοχή μου, στις δημοπρασίες του γάλακτος είχαμε μια αύξηση 2,5 πένες ανά λίτρο για το γάλα που πουλήθηκε. Και νομίζω μιλώ για περίπου στοιχεία. Άρα είναι τη συνολική τιμή 23,5, 23,5 πένες ανά λίτρο. Και το κόστος παραγωγής μου λένε είναι μεταξύ 24 και 25 πένες. Άρα δεν φτάσαμε σε κάλυψη του κόστους παραγωγής ακόμα και όλοι καλωσορίζουμε το γεγονός ότι οι τιμές αυξάνονται, διότι για να επιβιώσει ο τομέας πρέπει να παράγουν οι γαλακτοπαραγωγή με κέρδος, όχι με απώλεια. Στην περιοχή μου πολλοί παραγωγοί, επειδή έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα, ακόμα και σε αυτή την, ε, τιμή, για να εξυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, το, το κόστος είναι μεγάλο και ε, επειδή δεν τους πιέζουν οι τράπεζες επιβιώνουν. Μόνο έτσι επιβιώνουν. Εξαρτώνται κατά πολύ από την υποστήριξη των τραπεζών. Πρέπει να πω, η παρέμβαση δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση, όλοι το γνωρίζουμε και συμφωνούμε. Και όπως προανέφερα και είπα δημοσία, κανείς δεν θέλει να επιστρέψουμε στις παλιές μέρες των ε, λιμνών από γάλα και των βουνών από βούτυρο. Θα πρέπει να βρούμε καλύτερη λύση. Και ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στην Ευρώπη δεν ελέγχουμε το μέλλον. Εξαρτώμεθα από αυτά που θα γίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Εξαρτώμεθα από την ε, αποκατάσταση οικονομική ηρεμία στον κόσμο. Θέλουμε, εξαρτώμαστε από την Κίνα που θέλουμε να ξαναρχίσει εισαγωγές και εξαρτώμεθα και από αυτά που θα γίνουν και στη Νέα Ζηλανδία. Ε, πιστεύω λοιπόν, εφόσον δεν ήμασταν εξάρτητοι, ότι πρέπει να εξακολουθούμε να παρακολουθούμε προσεκτικά τι γίνεται. Δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από το πρόβλημα. Μέσω μακροπρόθεσμα μέτρα χρειάζονται, τα οποία μέτρα θα αποκαταστήσουν την, τον τομέα στην παλιά κατάσταση και θέλουμε να επιβιώσει το τομέα, διότι αν δεν έχουμε γαλακτοπαραγωγούς στην Ευρώπη, πού θα βρεθούμε. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους γαλακτοπαραγωγούς να μπουν στον τομέα και πρέπει να αποφασίσουμε εδώ ποιο είναι ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα προβλήματα διαφέρουν ακόμα και εντό ενό κράτου μέλου. Άκουσα τον Άλμπερ Ντε αυτά που είπε. Είπε μια ιδέα. Να αποσύρονται πιο νωρί οι παλιοί, οι ηλικιωμένοι παραγωγοί. Αν δεν εφαρμοστεί αυτό σε κάθε κράτο μέλο, ε, δεν ισότιμε συνθήκε. Κανεί δεν κερδίζει το τέλο ή μόνο μια μικρή περιφέρεια κερδίζει. Από αυτή την έποψη λοιπόν πρέπει να με πείσετε ότι ένα σύστημα ε, πρώιμης συνταξιοδότησης, απόσυρσης θα είναι ωφέλιμο. Ε, πρέπει να διαρωτηθούμε πρώτα γιατί η τιμή του γάλακτος που αποδίδεται στον παραγωγό είναι τόσο χαμηλή. Η τιμή που καταβάλλεται στον παραγωγό είναι χαμηλή και δεν ωφελήθηκε ο καταναλωτή, διότι ακούσαμε σήμερα το πρωί ανθρώπου να μα λένε ότι ο καταναλωτή εξακολουθεί να πληρώνει τιμέ που πλήρωνε πριν από 12, 18, 24 μήνε για το ίδιο λίτρο γάλα. Πού πήγαν τα χρήματα λοιπόν, πρέπει να ανακαλύψουμε. Ποιο τα πήρε τα χρήματα, ο παραγωγό δεν τα πήρε, ο καταναλωτή δεν τα πήρε. Άρα υπάρχει ένα κενό μεγάλο ανάμεσά του που πρέπει να ερευνηθεί. Σε πολύ ψηλό επίπεδο για να μάθουμε τι τρέχει, πού πήγαν τα χρήματα. Και όπως προανέφερα, διαφέρουν τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι ίσως βλέπουμε μία αμυδρή λάμψη ελπίδας. Αλλά δεν νομίζω ότι ξεφύγαμε από το δάσος ακόμα. Πρέπει να επικεντρωθούμε επί μέσω μακροπροθέσμων μέτρων, τα οποία θα εξασφαλίσουν το μέλλον του τομέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ James, Χριστίνα Μόρβεϊ. Ευχαριστώ. Σίγουρα η κύρια ερώτηση είναι η διαχείριση της κρίσης. Πέρα από αυτά τα μέτρα δηλαδή πρέπει να αναρωτηθούμε για την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να καταλάβει ότι χωρίς συγκεκριμένη ρύθμιση δεν οδηγούμεθα πουθενά. Δεν ε, υπάρχει μόνο η γεωργία που μπορεί να λειτουργήσει εφόσον η παραγωγή και οι αγορές δεν είναι ρυθμισμένες. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να το καταλάβει αυτό. Η άλλη μου ερώτηση έχει να κάνει με την οργάνωση των αγορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ρωτάω είναι έτοιμη να πει όχι στην παγκοσμιοποίηση έτσι όπως αυτή επιβάλλεται από τον ΠΟΕ είναι διατεθειμένη να πει όχι σε μια κατάσταση ακραίως φιλελεύθερη, όπου για παράδειγμα στη Βραζιλία εισαγάγουν σόγια σε τεράστιες ποσότητες, ενώ πολλές φορές είναι μολυσμένη η σόγια αυτή. Είναι κάτι που δημιουργεί δυσκολίες και στους Ευρωπαίους γεωργούς. Έχουμε μια κρίση. Πώς λοιπόν θα λυθεί το πρόβλημα λέμε, α, θα εξάγουμε γάλα σε σκόνη και θα το στείλουμε σε τρίτες χώρες, σε φτωχές χώρες, όπου η σκόνη αυτή η γάλακτος θα καταστρέψει τους ντόπιου παραγωγούς. Γιατί να μην υιοθετήσουμε τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της κρίσης κάποια έκτακτα μέτρα. Μέτρα επίσης χρειάζονται και στα διάφορα κράτη-μέλη. Ιδιαίτερα θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στην κατάσταση στις νέες χώρες-μέλη. Είναι γνωστό ότι οι αγορές μας τέθηκαν στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 100%. Και τι πήραμε ως αντάλλαγμα, ένα ελάχιστο κομμάτι ενίσχυση. Τουλάχιστον για τις χώρες αυτές λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πούμε πως τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της κρίσης θα έπρεπε να τους επιτρέπουμε να εισαγάγουν μέτρα προστασίας των αγορών τους. Γιατί βλέπουμε ότι το μόνο που γίνεται είναι ότι εξάγεται η κρίση προς τα εκεί. Στην Ουγγαρία εισαγάγουμε γάλα που έρχεται από το εξωτερικό, σπάει τις τιμές στην Ουγγαρία, καταστρέφει τους ε, Ούγγρους αγρότες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί μια τέτοια κατάσταση λοιπόν, είναι αδύνατον. Η ε, διατροφική αυτάρκη, δηλαδή το πρώτο στοιχείο για να είμαστε αυτάρκης, είναι πολύ βασικό και το κυριότερο γι' αυτό είναι να μπορούν οι ίδιοι οι παραγωγοί και αγρότες να αποφασίζουν τι θέλουν να παράγουν, ώστε να μπορούν να στηρίξουν τη δικιά τους την αγορά και να μην υποχρεώνονται να εισάγουν παρά μόνο εφόσον πραγματικά χρειάζονται την ε, εισαγωγή αυτή κάποιου προϊόντος. Πάρα πολλοί γεωργοί πραγματικά βρίσκονται στα όρια της αυτοκτονίας. Υπάρχουν αγρότες που έχουν καταστραφεί οικονομικά τελείω. Η ύπεθρος επίση καταστρέφεται. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση λοιπόν. Πρέπει να ληφθούν μέτρα οπωσδήποτε. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο που τηρήσατε μεγάλο ε, ενθουσιασμό. Το συζητάτε με ενθουσιασμό αυτό το θέμα. Αλλά πρέπει να χειριστούμε σωστά το χρόνο, αλλιώ θα μιλάμε όλο το απόγευμα μόνο για το γάλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το χρόνο που προσφέρετε στην Επιτροπή μας ως Πρόεδρος για να συζητήσει το θέμα του κλάδου αυτού. Πρώτα απ' όλα, όπως και συνάδελφος από την Βόρεια Ιρλανδία, και εγώ θέλω εδώ πέρα να ρωτήσω μερικά πράγματα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που λέει ότι οι τιμές του γαλακτομικού παρέα στην τομέα 20% αυξήθηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία από τον Ιούνιο ε, φέτος και μετά. Ωραία, μακάρι να ήταν έτσι, αλλά όπως είπε και ο Νίκολσον, οι τιμές αυτές δεν έχουν φτάσει ακόμα και θέλω να επενθυμίσω επίσης στην Επιτροπή ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή στη χρονιά όπου οι τιμές είναι χαμηλές στο χαμηλότερο επίπεδο. 15 με 16 πένες το λίτρο. Πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά τα ποσά, αυτά τα στοιχεία. Θα ρίνουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δουλέψει σοβαρά και να φροντίσει η γαλακτοπαραγωγή και οι αγρότες να έχουν μια σταθερή αγορά. Δεν είναι δυνατόν να ξαναβρεθούμε στη, στα πάνω και κάτω αυτά 2007-2009. Όχι, πρέπει να υπάρχει κάτι σταθερό στο γαλακτοκομικό τομέα για να μπορούν να βασίζονται στο μέλλον οι αγρότες αυτοί και όχι να εξαφανίζονται οι νέοι αγρότες, οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Θέλω επίση να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει και πώς μπορεί να κρατηθεί η τιμή σταθερή. Μας είπαν ότι θα κοιτάξουν να βρουν μια τεχνικού είδου λύση όσον αφορά τη συζήτηση για τα GM. Θέλω λοιπόν να τους ζητήσω όσο γίνεται πιο γρήγορα και καλύτερα γρήγορα παρά αργότερα να μας δώσουν κάποια απάντηση. Μάρκ Ταραμπέλα έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Δύο λόγια έχω να πω. Ρύθμιση. Είναι αναγκαία ρύθμιση στον τομέα αυτό, που υπάρχει κρίση στην ε, προσφορά. Είχαμε τη θέση που το 2003, αλλά βέβαια υπάρχουν εξελίξεις. Έχει αλλάξει η κατάσταση επιγής. Είχαμε τη δημοσιονομική κρίση, την οικονομική κρίση, τη γαλακτοκομική τώρα, την κρίση στην ε, προσφορά. Ναι, γίνονται κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να μιλάμε για ρύθμιση. Είμαι λοιπόν από τους λίγους που δεν ψήφισα τελικά το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, γιατί όλες οι τροπολογίες που πηγαίνανε προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής ρύθμισης, ακόμα και οι ελάχιστες που θέλανε να παγώσει το ποσοστό των ποσοστώσεων ε, προσωρινά, δεν υιοθετήθηκαν. Οπότε τελικά η ρύθμιση δεν είναι το κύριο στοιχείο. Γι' αυτό και προτίμησα να κρατήσω θέση αποχής. Σε επίπεδο συμβουλίου τώρα. Η Ιταλία, η Πολωνία, για παράδειγμα, είναι χώρες που σίγουρα βαραίνουν. Λοιπόν, θα σας πω δύο σημεία. Τη δήλωση εκεί που συμφωνούν οι 20 χώρες προς το παρόν, που μιλάνε για νέους τρόπους ρύθμισης. Είναι γραμμένο και μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες. Δήλωση των ηγετών κρατών και κυβερνήσεων που λέει ότι να μην βαζόμαστε μόνο στους κανόνες αγοράς, αλλά είμαστε σε θέση και να ανταποκριθούμε σε αυτούς. Σε κάποιο σημείο άλλο λέει ότι πρέπει να δούμε τα, μέσα τα οποία μας βοηθούν να διαχειριστούμε την αγορά σήμερα, να είναι πιο ελαστικά, πιο αποτελεσματικά, ε, όσον αφορά την αστάθεια που επικρατεί στις τιμές μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, για να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα πλαίσιο, και το Συμβούλιο της Δευτέρας ήταν ε, βασικό, πρέπει να πω ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την Κομισιόν, γιατί μετά από τις δηλώσεις της κυρίας Φίσελμπουλ που ήρθε και είπε ότι έχει καλά νέα στις 15 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο και μας εξέφρασε την επιθυμία της ε, τα μέτρα μηνυμής να είναι 15.000 ευρώ το όριο, εγώ συζήτησα με τον Περιφερειακό Υπουργό μου, τον κύριο Λουτγέν, ο οποίος μου είπε ότι χτες πήρε το σημείο με αυτό και δεν έχω βέβαια περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στους γαλακταπαραγωγούς και τους υπόλοιπους αγρότες. Δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν αφορούν μόνο τους γαλακτοπαραγωγούς, αφορούν όλους τους αγρότες. Ε, τελικά ελάχιστα θα πάρουν. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Εμείς αλλιώς είχαμε καταλάβει την πρόταση της Επιτρόπου. Οπότε πρέπει να δούμε, εμείς η Επιτροπή μας δηλαδή, πώς η Εκτελεστική Επιτροπή σκοπεύει να εφαρμόσει το μέτρο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα την Επιτροπή πριν. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μάρτιν Χάουσλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως πράσινοι καταψηφίσαμε το ψήφισμα, διότι θεωρούμε ότι αποφεύγει τα βασικά θέματα, δηλαδή κυρίως την υπερπαραγωγή, την πλονάζουσα παραγωγή. Και βρίσκω και απογοητευτική την απάντηση της Κομισιόν. Αυτό που κάνει η Κομισιόν είναι κάπως ε, σαν κάποιος που ε, περπατάει μέσα στο δάσος νύχτα και τραγουδάει για να δώσει θάρρος στον εαυτό του. Στην πραγματικότητα οι λόγοι είναι εποχιακοί, που κινητοποιούνται δηλαδή και είναι και γιατί υπήρξαν οι κινητοποιήσεις. Αντίθετα με αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχουν αλλαγές τάσεων στην αγορά. Θα προτιμούσα να είχε πει και λίγο περισσότερα νούμερα. Δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση της αγοράς. Πού βρίσκεται η πλεονασματική, σε ποιο ύψος πλεονασματική παραγωγή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με ενδιαφέρει επίσης εάν η πολιτική εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πραγματικά έτσι όπως μας την περιγράφουν και αν δεν πλήττει πραγματικά χώρες του τρίτου κόσμου. Σε ποιες χώρες κατευθύνθηκαν αυτές οι εξαγωγές, οι επιδοτούμενες εξαγωγές και υπάρχουν κάποιες χώρες που η αγορά τους επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο και όπου ενδεχομένως σε χωριστή του κόσμου προκαλούμε πραγματικές καταστροφές στις αγορές τους με τις επιδοτούμενες εξαγωγές μας. Επίσης δεν άκουσα αυτό που ανακοίνωσε μεν η Επίτροπος και συμφωνήσαμε εμείς, δηλαδή ότι θα αναλυθούν πρωτοβουλίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενισχυθεί η θέση των γαρακτοπαραγωγών. Διότι ναι μεν το συζητούμε αυτά, τα συζητούμε αυτά, αλλά ποιου μηχανισμού θα προσφέρουμε στους ε, γαλακτοπαραγωγούς για να μπορέσουν να ενισχύσουν την θέση του στην αγορά. Δηλαδή, εν τέλει, με λίγα λόγια, εγώ δεν βλέπω λύση για την κρίση. Πολλοί γαλακτοπαραγωγοί ακόμα παλεύουν για να εξασφαλίσουν το αύριο και δεν ξέρω πώ θα τα καταφέρουν. Έχω την εντύπωση ότι από πλευρά Κομισιόν και Συμβουλίου δεν πράττουν τίποτα. Κάθονται με τα χέρια σταυρωμένα και περιμένουν απλώ να Λήξη η κρίση. Σας ευχαριστώ Μάρτιν. Ζωζέ Μποβέ. Δύο λεπτά. Νομίζω ότι όσο ακούσαμε από την Κομισιόν πριν από λίγο δεν είναι αξιοπρεπή, δεν είναι άξια της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας σήμερα. Είχαμε την ε, περιά του γάλακτος μέχρι 5 Οκτωβρίου σταματάει. Αν 5 Οκτωβρίου δεν υπάρξει πραγματική απάντηση αυτό που περιμένουν όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες τα πράγματα θα πάνε πολύ πιο άσχημα, γιατί οι παραγωγοί δεν θα έχουν πια καμία ελπίδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό, αλλά όχι μόνο και τα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό και εδώ χαιρετίζω το διάβημα της Γαλλίας μαζί με τη Γερμανία, που βρήκαν σύμφωνε και άλλε 18 χώρε. Συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν και στρέφομαι προς την Επιτροπή γιατί σήμερα έχετε μέσα στη διάθεσή σας. Τα σημερινά μέσα λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Παραδείγματα. Σήμερα πρέπει ξεκάθαρα να χρησιμοποιηθούν οι προσωρινές ενισχύσεις στην εθελοντική μείωση των ποσοστώσεων. Έγινε τη δεκαετία του 90, υπάρχει το μέσον. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι σούπερ εισφορές ε, ποινής για να συμπληρωθεί ο φάκελος, για να μειωθεί ο όγκος, αντί να υπάρξει χρηματοδότηση της εξαφάνισης των αγροτών, να το στέλνουμε στη σύνταξη. Να κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Επίσης, χρειάζονται κυρώσεις και έχετε τα μέσα να το κάνετε στις ποσοστώσεις που συνεχίζουν να παράγονται ενώ έχουν πουληθεί σε αγρότες. Αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες. Έτσι καταστρέφεται η δυνατότητα διαχείρισης που έχει κάθε χώρα. Απαράδεκτο. Έπειτα πρέπει να εμποδίσουμε την παραγωγή υπερβολικών ποσοστήτων στο τέλος μιας περίοδου. Έχουμε τα μέσα να το κάνουμε και αυτό, γιατί αυτό αποσταθεροποιεί τις αγορές. Και τέλος να υποφεληθούμε από όλες αυτές τις δυνατότητες, ώστε να προσφέρουμε και πάλι ισορροπία στον όγκο των προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν είναι δυνατόν ορισμένε χώρε να αναγκάζονται να εισάγουν όπω είναι η Ιταλία, η Ισπανία και οι 12 χώρε που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα. Πρέπει να υποφεληθούμε λοιπόν από αυτή την κατάσταση για να επιφέρουμε εκ νέου ισορροπία στην παραγωγή. Αν δεν υπάρξει αυτή η ισορροπία στην παραγωγή, δεν θα βγούμε από την κρίση. Έχετε στη διάθεσή σας μέσα σήμερα, πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε. Πέντε χρόνια έχουμε ακόμα στο σημερινό καθεστώς ποσοστώσεων. Μην κάνουμε σαν να μην έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας, τα έχουμε. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ράσμουσεν για την παρουσίασή του. Ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα στατιστικά και θα ήθελα να τα παραλαμβάνουμε αυτά επί τακτικής βάσης. πρόθεσμα, θεωρούσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είχαν απόλυτο δίκαιο στις προτάσεις τους. Θεωρούσα ότι η χρήση των, της πανέβασης όπως έλαβε χώρα ήταν σωστό εργαλείο, σωστή χρήση των υφισταμένων εργαλείων. Αλλά θέλω να παροτρύνω και το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρησιμοποιούν πιο ουσιαστικές αντιδράσεις για αυτή την κατάσταση διότι αυτό θα ήταν μια λύση για κατεπήγον πρόβλημα και νομίζω ότι σωστά ο κύριος Ράσμουσεν είπε ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστούν τα μακροπρόθεσμα διαθετικά προβλήματα του τομέα. Το σημαντικότερο θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι ο δυσλειτουργικός μηχανισμός διαμορφώσεως των τιμών αγοράς. Δεν υπάρχει σαφής διασύνδεση μεταξύ τιμής ή αξίας στο λιανεμπόριο και τιμής που ε, εμφανίζεται στην πλευρά της ε, προμήθειας ε, του παραγωγού. Δύσκολο πρόβλημα. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας γενικός δεντολογικός κώδικας. Δύσκολο. Αλλά δεν μπορείτε να θεσπίσετε νομοθεσία για καθορισμό περιθωρίων εντός του τομέα. Αυτό δεν θα βοηθούσε καθόλου. Και αυτό που είναι πιο ξεκάθαρο είναι ότι η μεγαλύτερη επιρροή διαμορφώσεως των τιμών που είναι παραγωγός είναι η παγκόσμια τιμή και οι παγκόσμιες τιμές των βασικών γεωργικών προϊόντων πρόσφατα συνδέονται με τις παγκόσμιες τιμές, κυρίως οι τιμές βασικών προϊόντων στον ενεργειακό τομέα. Άρα οι τιμές έγιναν πολύ πτυτικές. Δεν το είδαμε αυτό μόνο στο γάλα, αλλά και στο σιτάρι και σε άλλα αγροτικά βασικά προϊόντα. Η άμεση αντίδραση που προανέφερα και που ακούγεται εδώ μυρίζει από προστατευτισμό. Και θα πω εδώ αυτό που λέει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προστατευτισμό δεν είναι ποτέ η απάντηση, δεν είναι απάντηση εν συγκρίση με τον ανταγωνισμό. Και υποστηρίζω την κατάργηση των ρυθμιστικών μηχανισμών της αγοράς, όπως οι ποσοστώσεις, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι γίνεται πιο μακροπρόθεσμα. Η πτητικότητα έδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο γεωργικό τομέα, διότι είναι μακροπρόθεσμες οι επενδύσεις μας Οπότε θα χρειάζεται μακροπρόθεσμο σύστημα παρεμβάσεων σαν κομμάτι της προτάσεως που θα υποβληθεί στον ΠΟΕ. Αυτά και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελάνς έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ πολύ. Χθε το βράδυ μίλησα με μία φίλη η οποία πήγε στο Αφγανιστάν και μετά στη Βοσνία και μιλούσαμε για τους τρεις μεγάλους παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα στον κόσμο, που είναι το νερό, η ενέργεια και τα τρόφιμα. Και εμείς τι κάνουμε στην Ευρώπη, δυσκολεύουμε την ζωή των αγροτών μας. Ενώ εκεί ακριβώς είναι ένα από τα κύρια προβλήματα του κόσμου. Δεν είμαι κάποιος που δεν παρακολούθησα την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την άκουσα, άκουσα τις λύσεις που προτείνει και που δεν είναι μόνο η προσφορά. Συμφωνώ και είχαμε και τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε τη συζήτηση αυτή να τη διευρύνουμε περισσότερο και να μην συζητάμε μόνο όταν πρόκειται να ψηφίσουμε. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολύ λίγα. Ωραία με το αποκορυφωμένο γάλα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό που με απασχολεί εμένα πολύ περισσότερο όμως είναι η απόλυτη ησυχία που ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το μακροπρόθεσμο στάδιο. Τι θα κάνουμε αργότερα. Γιατί εντάξει, μιλάμε τι θα κάνουμε τώρα με τι επιστροφέ από τι εξαγωγέ. Ναι, αλλά μακροπρόθεσμα. Εγώ πιστεύω ότι ο τομέα μα ε, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά λύση με αυτό το σύστημα των επιστροφών ε, σε εξαγωγέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά τι κάνει. Ε, τα ίδια της τα προϊόντα δεν τα πληρώνει όσο θα έπρεπε. Μακροπρόθεσμα λοιπόν, τι θα γίνει. Συμφωνώ με την Επιτροπή ότι και η αγορά πρέπει να κάνει τη δικιά της τη δουλειά, αλλά δεν φτάνει. Γιατί όταν η αγορά οδηγεί σε πολύ ψηλά επίπεδα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εμεί αυτά τα ακραία φαινόμενα πρέπει να τα περιορίζουμε. Εντάξει την αγορά να τη δούμε, το έχω πει πολλέ φορέ. Και συμφωνώ, ναι, και έκανα και την έρευνα για τις αγορές. Κοιτάξτε, να, σε Ολλανδική εφημερίδα, και εδώ δεν μιλάω για μια αγροτική, μια μεγάλη Ολλανδική εφημερίδα, ξεκινάει να ε, κάνει διαφημίσεις από παραγωγούς ε, γαλακτοκομικών προϊόντων οι οποίοι αρχίζουν και λένε εμείς δεν συμφωνούμε με τα σούπερ μάρκετ γιατί μας πληρώνουν πάρα πολύ λίγο. Και έτσι δεν μπορούμε εμείς να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή. Να λοιπόν, ότι με τα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν να ζήσουν οι αγρότες. Και οι στάνταρτ επίσης. Κάτι λοιπόν σημαίνουν όλα αυτά. Τα δύο τελευταία. Πρώτον, η συζήτηση για το τι θα γίνει μακροπρόθεσμα επίσης πρέπει να, πρέπει να γίνει. Γιατί οι αγρότες θέλουν ε, φυσικά να εξασφαλίσουν προϊόντα για την αγορά, πολύ ωραία, αλλά κάπως πρέπει να στηρίζονται και αυτοί. Και τέλος, επενδύσεις χρειάζονται και όσον αφορά την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Το λέμε, αλλά δεν μας ακούει κανείς. Και στο γαλακτοκομικό τομέα ισχύει αυτό. Γιατί και εδώ υπάρχουν ευθύνε για τη θέρμανση του κλίματος. Λοιπόν, πώς θα διορθωθεί η κατάσταση. Χρειάζονται επενδύσεις. Να γίνουν. Γιατί θα βοηθήσουν όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και θα βοηθήσουν στην εικόνα που έχει αγροτικό τομέα. Ρωτάω λοιπόν την Επιτροπή Τάξη, σκεφτεί αυτά και τι απάντηση έχει να μου δώσει. Συμφωνούμε όλοι επ' αυτού. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις κλιματολογικές αλλαγές έχει μια θέση απόλυτα ομοιομορφή. Η κυρία Ματιού έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξεπλάγει όταν άκουσα αυτά που μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω την εντύπωση ότι ο κύριο Ράσμουσεν αυτή τη στιγμή ε, δεν έχει πατήσει πόδι πρόσφατα στι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Την πράσινη εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα την πέρασα με το Συνδικάτα των Γεωργών τη περιοχή μου, επανειλημμένα του συνάντησα και πήγα στι εκμεταλλεύσεις των γαλακτοπαραγωγών και κύριε Ράσμουσεν, αν πηγαίνατε να μιλήσετε εκεί και να τα πείτε αυτά στου γεωργού, σα διαβεβαιώ ότι θα υπήρχαν πολύ βίαιε αντιδράσεις, διότι του λέτε ότι όλα πάνε καλά και ότι η τιμή του γάλατο αυξάνεται από τον Ιούνιο, είναι σαν να του κοροϊδεύετε και σα διαβεβαιώ ότι σχεδόν μα κοροϊδεύετε και εμά εδώ, λέγοντα ότι όλα πάνε καλά. Εγώ έτσι αισθάνθηκα και δεν είμαι ικανοποιημένη. Πάει άσχημα ο τομέα, δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντιδρά αρκετά στα όσα λέει το Κοινοβούλιο και οι Υπουργοί. Το να λέτε αυτά δεν είναι πολύ εντάξει απέναντί μας. Θα ήθελα να πω όμως ότι υπάρχουν κάποια μέτρα που ελήφθησαν. Είναι καλό το ότι συνεδριάζει το Συμβούλιο υπό την πίεση κάποιων υπουργών και ελπίζω ότι τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν επί τη ευκαιρία του εκτάκτου Συμβουλίου θα καθησυχάσουν τον αγροτικό κόσμο διότι ο αγροτικός κόσμος το χρειάζεται, ε, απελπισμένος είναι, υποφέρει ανεξάρτητα από τα μέτρα που ελήφθησαν Ελπίζω, όπως είπαν και συνάδελφοι, ότι τελικά τα μέτρα που θα ληφθούν θα έχουν αποτέλεσμα. Είναι ένα επάγγελμα η σειρά ετών με τις διάφορες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ δεν έχει μακροπρόθεσμο όραμα όσον αφορά το επάγγελμά του. Είναι ένα επάγγελμα που έγινε πάρα πολύ αγχωτικό, είναι σε δυσχερή θέση, κυρίω για του ε, νέου και διάφορε αναδιαρθρώσει που προβλέπονται δεν, και προβλέφθηκαν και εφαρμόστηκαν δεν τους επιτρέπουν να έχουν μακροπρόθεσμο όραμα. Αυτή η κρίση του γάλακτος, το τέλος των ποσοστώσεων ήταν μεγάλο σφάλμα και ελπίζω ότι θα προβλεφθεί ένα σύστημα ρύθμισης που θα εναντάξει το ονοματό του. Διότι όπως είπε η κυρία Ντελάγκε, δεν βλέπω πώς σήμερα μπορούμε να περάσουμε από ένα σύστημα ρύθμισης Πώ θα τα κάνουμε χωρί ένα σύστημα ρύθμιση. Μπορεί να μην το λέμε ποσοστώσει πλέον, αλλά πρέπει να ελέγξουμε την γαλακτοκομική παραγωγή, την παραγωγή γάλακτο. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συνάψεω συμβάσεων μεταξύ παραγωγών και βιομηχανία και να μην λησμονούμε και του μεταποιητέ και του παραγωγού. Υπάρχουν θέσει απασχόληση που είναι πάρα πολύ σημαντικέ σε αυτό το τομέα και στη βιομηχανία και στη μεταποίηση. Και και εξίσου υπάρχουν και σημαντικέ θέσει, αριθμό θέσεων και για την καλλιέργεια. Για του καλλιεργητέ μα, μάλλον του παραγωγού μα. Ο Πίτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία σχόλια έχω όσον αφορά αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, οι τάσει των ε, τιμών. Αυτά που είπατε είναι σωστά, αλλά θυμηθείτε ότι δεν καλύπτονται, δεν καλύπτεται το κόστος παραγωγής. Όλα όσα έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σταθεροποιήσει την αγορά ή ό,τι θα κάνει πρέπει αυτό να το έχει υπόψη της. Θα ήταν εσφαλμένο να χαλάσουμε αυτό που, να ανοίξουμε αυτά που έχουμε στην παρέμβαση. Όσον αφορά την εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές στην αγορά αυτή, πρέπει να γίνει από πλευράς προμήθειας κάτι. Μάλλον διατροφής να γίνει κάτι. Να χρησιμοποιούνται τα σωστά τυριά, στο μαγείρεμα, να χρησιμοποιήσετε τα σωστά συστατικά. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα στην εσωτερική αγορά για να προωθήσουμε τη χρήση των σωστών προϊόντων. Μακροπρόθεσμα. Χρειαζόμαστε νέες συμφωνίες, συμβάσεις μεταξύ των παραγωγών και του τομέα του εμπορίου. Όσον αφορά τη Γερμανία, δεν θα μπορούσα να πω ότι το εμπόριο είναι εχθρός του παραγωγού. Το εμπόριο βοηθά τους παραγωγούς. Θα πρέπει να προσέξουμε τα δικαιώματα των παραγωγών και να τα ενισχύσουμε. Για να μην είναι α... άνευ υπεράσπιση, η παραγωγή. Λοιπόν, και θα πρέπει να μπορούμε να καλύψουμε το κόστος της παραγωγής. Εντάξει, δύο λεπτά ακριβώς λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, George Lyon. Ε, Έχει το λόγο για δύο λεπτά. Θα είμαι σύντομος Πρόεδρε. Καταλαβαίνω ακριβώς ότι δεν περισσεύει ο χρόνος. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι καλωσορίζω μεν την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα πρέπει δε να είμαστε πολύ προσεκτικοί μπορεί οι ιονοί να δείχνουν ότι υπάρχει ανάκαψη αγοράς όσον αφορά τους γαλακτοπαραγωγούς θα περάσει χρόνος αρκετός για να ωφεληθούν και να έχουν κέρδη αυτοί που έχουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις και να έχουν καλύτερα κέρδη ως παραγωγή. Θα ήθελα να θέσω ένα συγκεκριμένο θέμα τις συζητήσεις που είχαμε με τον Γάλλο Υπουργό το πρωί. Εκεί ο Γάλλος Υπουργός έκανε κάποιες προτάσεις. Πολλές από τις προτάσεις ε, μου δημιουργούσαν πρόβλημα. Αλλά σε κάποιο τομέα αναφέρθηκε που νομίζω ότι σαν Επιτροπή και σαν Κοινοβούλιο θα πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα. Διαφάνεια της όλης αλυσίδας της τροφικής του γάλακτος στη Γαλλία έγινε μια βασική ανάλυση της αλυσίδας αυτής και ό,τι εκπλήξεως το κέρδος δεν το παίρνουν οι παραγωγοί. Και ό,τι εκπλήξεως ούτε οι περαγορές ε, παίρναν τα κέρδη, αλλά ε, κέρδη οι μεταποιητές έβγαζαν τα περισσότερα. Αυτά δείχνει η μελέτη που έκαναν οι Γάλλοι όσον αφορά την αγορά γάλακτος. Οπότε επιστρέφουμε στο πρόβλημα. Δηλαδή, και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές πέφτουν θύματα μιας αγοράς που δεν λειτουργεί. Δεν αντικατοπτρίζει τις πτώσεις των τιμών στην παραγωγή και όταν είναι καλύτερος ο καιρός δεν επιστρέφουν τα κέρδη στους παραγωγούς. Οι Γάλλοι πρότειναν ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε τα, στις συμβάσεις μακράς διαρκείας που θα επιτρέπουν αυτές οι αλλαγές των τιμών να αντικατοπτρίζονται στον παραγωγό και όλοι στην αλυσίδα της παραγωγής να αμείβονται δίκαια. Αυτό πρέπει να το συζητήσει το Κοινοβούλιο. Περιμένουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα εξετάζει τι γίνεται με την τροφική αυτή αλυσίδα σε όλη την Ευρώπη και είπε η κυρία Φίσορμπολ Μπόλ το Δεκέμβριο θα υποβληθεί η έκθεση και θα πρέπει να πιέσουμε ούτω ώστε να έχουμε ένα σύστημα που να λειτουργεί και για του καταναλωτέ και του παραγωγού. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ακολουθήσει πολιτική που θα στέφεται και την αγορά, η αγορά πρέπει να λειτουργεί και για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές. Και αυτό είναι κάτι που το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσει πάρα πολύ και να ασκήσει τις δύο πίεσει. Ευχαριστώ, Τζόρτζ. Σι Κυριέσκη. Σας ευχαριστώ. Ήταν ενδιαφέρουσα η παρέμβαση αυτή. στην πραγματικότητα αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι δεν δραστηριοποιούνται τα όργανα. Και βλέπω τελικά τους γεωργούς να στρέφονται σιγά σιγά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό δεν υπήρξε επαρκής εποπτεία, γιατί έγινε αυτό. Πόσοι αγρότες έχουν εγκαταλείψει τη δραστηριότητά τους. Πού βρίσκονται οι αιτίε Έχει μειωθεί η ζήτηση λόγω κρίσεως. Υπάρχουν άλλες αιτίε για την κρίση που παρατηρείται στο γαλακτοκομικό τομέα. Αυτό είναι το ερώτημα. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να προαγάγει κανείς, να προαγάγουμε δηλαδή εμείς όλοι και κάποιο όραμα να διευκρινίσουμε τι επιθυμούμε. Η θα απολέσουμε παν ίχνος αξιοπιστίας στα μάτια των Γιώργων. Ακούμε διαρκώς ότι το τάδε υψηλό ποσοστό δαπανάται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για την κοινή αγροτική πολιτική. Μα πού πηγαίνει. Στεφάν Λεφόλ, τελευταία παρέμβαση. Θα είμαι σύντομος, γιατί έχουν υποθεί λίγο πολύ όλα. Η κρίση αυτή δεν έχει να κάνει ειδικά με το γάλα. Είναι μια γενικότερη κλίση. Είναι συγκυριακή, είναι η μείωση των τιμών και χρειάζονται συγκυριακά μέτρα. Και εδώ όσον αφορά τον έλεγχο της προσφοράς, συμφωνώ με τον Ζωζέ Μποβέ, ότι πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη μέτρα, ώστε να μην μπαίνει παραγωγή στην αγορά υπερβολικά μεγάλη, με αποτέλεσμα μετά να πρέπει να την αποσύρουμε ε, στην παρέμβαση. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Δεύτερο, θα καταφέρουμε να ηρεμήσουμε το θυμό των αγροτών, ο οποίος, προσοχή, δεν θα περιοριστεί στους γαλακτοπαραγωγούς, αλλά θα μπορέσουν να ηρεμήσουμε το θυμό τους μόνο αν μπορέσουμε να δώσουμε μια ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Γιατί αυτό ακριβώ είναι που λείπει σήμερα. Και εδώ ερχόμαστε στο θέμα της ρύθμισης. Πώς δηλαδή διαχειριζόμαστε τη γεωργία και τα τρόφιμα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί δεν είναι δυνατόν να κάνουμε όπως κάναμε και παλιά. Το θέμα του ελέγχου της προσφοράς κανένας δεν έχει καθίσει να βάλει μια εναλλακτική λύση επιτάπητος. Κανείς. Και σας το λέω ξεκάθαρα. Όταν δεν θα ελέγχεται από την Ευρώπη η προσφορά, θα έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Και η αγορά ένα πράγμα θα ρυθμίσει μόνο θα δώσει μεγαλύτερο κέρδος στους πιο ανταγωνιστικούς. Τελεία, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Η συζήτηση που γίνεται είναι πολιτική για τη ρύθμιση των αγορών και αφορά όλη τη γεωργία και τα τρόφιμα. Ωραία. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Ευχαριστώ βεβαίως και τον κύριο Ρασμούσεν που ελπίζω ότι στην έκθεσή του, στην αναφορά του θα μπορεί να, λάβει υπόψη πόσο δυσαρέσκεια υπάρχει στην Επιτροπή μας από αυτά που άκουσε συζήτηση για το γάλα ότι ελπίζουμε και ευχόμαστε οι πρωτοβουλίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι πρωτοβουλίε όλου του Κοινοβουλίου να εισακουστούν και σε συναντήσει της 5ης και τη 29 η και τη ε, 30 η Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, η δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου στον αγροτικό τομέα. Καλωσορίζω το Διευθυντή του Ελεκτικού Συνεδρίου, Edward Φένεση, της πρώτης ομάδας που είναι η Γεωργία και Φυσική Πόρη, ο οποίος μπορεί να μας παρουσιάσει τη γενική μεθοδολογία του Ελεκτικού Συνεδρίου για τον γαλακτοκομικό τομέα και ποια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα με τα πρόσφατα αποτελέσματα. Δώσω το λόγο στον Διευθυντή, τον κύριο Φένεση. Ε, ελπίζω να μπορέσει να μας κάνει μια παρουσίαση που θα κρατήσει περίπου 15 λεπτά, άντε 20 το πολύ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα εδώ εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε εσάς που μου επιτρέπετε να έρθω εδώ σήμερα και να σας παρουσιάσω το έργο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πιέζει, γι' αυτό θα προσπαθήσω κι εγώ να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος και περιττώ να σας πω ότι εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις μετά ευχαρίστως θα είμαι στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω. Πρώτα λοιπόν, να σας πω ότι αποτελείται από τέσσερις ομάδες ελέγχου το λεκτικό συνέδριο, ιδιαίτερα στους τομείς των δαπανών και υπάρχει και μία οριζόντια ομάδα ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου αριθμός 1 που εγώ θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των δαπανών που έχουν να κάνουν με την γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αλία, επίσης περιβάλλον, υγεία και προστασία του καταναλωτή έχει συνολικά περίπου 140 ελεκτές προσωπικό και συναφές και έναν προπολογισμό της τάξης του 58 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σύντομα, τώρα θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τη μεθοδολογία μας. Το ελεγκτικό συνέδριο εφαρμόζει τις διεθνείς προδιαγραφές ε, οικονομικού ελέγχου από την Ιντοσάι που είναι η Διεθνής Οργάνωση Ελέγχου Οργανισμών και τη ΑΕΦΑΚ επίσης που είναι η Διεθνής Ομοσπονδία για Ελέγχους ε, Οικονομικούς. Συμμετέχει επίσης ε, στην εκπόνηση των προδιαγραφών αυτών. Οι ευθύνε του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ο οικονομικός έλεγχος, ο έλεγχος της ε, αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την οικονομική διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δρούμε ως ανεξάρτητος ε, φύλακας των οικονομικών συμφερόντων και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, πολύ σύντομα θα σας ε, σχεγραφίσω κάπως τη μεθοδολογία του λεκτικού συνεδρίου, τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου και θα αναφερθώ λιγάκι και στη συνέχεια και στη δουλειά που κάνουμε όσον αφορά τον έλεγχο της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Γενικότερα μιλώντας λοιπόν, ο οικονομικός έλεγχος εξετάζει κατά πόσο οι οικονομικές συναλλαγές καταγράφονται ορθά και κατά πόσο είναι νόμιμα και νομότυπα εκτελεσμένες. Ο έλεγχος ε, που κάνει λοιπόν το λεκτικό συνέδριο βασίζεται στην ε, ετήσια δήλωση αξιοπιστίας, DAS, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, που ετησίως παρουσιάζει το ηλεκτρικό συνέδριο ε, στις αρμόδιες για τα δημοσιονομικά αρχές. Και έχουμε βέβαια και την διαδικασία απαλλαγής κάθε χρόνο. Για το 2008 η έκθεσή μα θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Ολομέλεια βέβαια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο. Όσον αφορά τη δήλωση αξιοπιστίας, αποτελείται από δύο ιδιαίτερα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα είναι η αξιοπιστία των λογαριασμών. Και το δεύτερο είναι γνωμοδότησή μας όσον αφορά την, ε, την ε, νομιμότητα και το νομότυπο των ε, συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι εξολογούμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πώς έχουν διαχειριστεί τα ποσά του προπολογισμού που τους αναλογούν, αν έχει γίνει σωστή διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη και Αξιολογούμε επίσης κατά πόσο οι οικονομικές συναλλαγές, έτσι όπως αναφέρονται στου λογαριασμού έχουν καταγραφεί σωστά και έχουν εκτελεστεί νόμιμα και νομότυπα. Με την πάροδο των ετών, το λεκτικό συνέδριο έχει κερδίσει όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών, παρόλο που μερικές φορές σε ορισμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Μέχρι τώρα πάντως η άποψή του όσον αφορά την νομιμότητα και τον ομότυπο των συναλλαγών ήταν αρνητική. Όσον αφορά την γεωργία, η δήλωση εξοπιστίας έχει δείξει ότι υπάρχει μια βελτίωση τα τελευταία χρόνια, κυρίως ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε το σύστημα AIAX και πολύ πρόσφατα επειδή χρησιμοποιούμε το σύστημα ενιαίων πληρωμών και ενιαίας περιοχής πληρωμών. Ακριβώς επειδή αυτά τα προγράμματα είναι πολύ σημαντικά, έχει δώσει πολλά χρήματα ε, το ελεγκτικό συνέδριο για αυτού του είδους τους ελέγχους τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να επαληθεύει την δαπάνη των χρημάτων βάση των δικαιούχων. Με την εισαγωγή αυτών των τελευταίων προγραμμάτων, η περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται κάποια παράνομη δραστηριότητα ή παράτυπη, οι περιπτώσεις αυτές έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχει μεγάλο, μεγάλη πιθανότητα σφάλματος και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι αγρότες πρέπει να τηρούν ιδιαίτερα περίπλοκους κανόνες και διατυπώσεις. Τώρα για τις λεπτομέρειες πώς το ελεγκτικό συνέδριο ετοιμάζει τη δήλωση αξιοπιστίας του δεν θα σας ε, το πω αυτό. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι γίνονται δοκιμές, ανάλυση συστημάτων προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι σωστά και κατά πόσο είναι αξιόπιστα. Το ελεκτικό συνέδριο επίσης χρησιμοποιεί και άλλες πηγές, δευτερογενείς αυτές, όπως είναι οι δηλώσεις των διαφόρων ε, σωμάτων που συμμετέχουν, των διαφόρων πλευρών, όπως είναι οι δηλώσεις των διευθυντών, των ε, οργανισμών που κάνουν τις πληρωμές, των ε, γενικών διευθυντών, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας κλπ. Επίσης, εφόσον μπορούμε και ανταποκρίνονται στα κριτήριά μας, χρησιμοποιούμε και τη δουλειά που κάνουν άλλοι ελεγκτές. Συνολικά λοιπόν όσον αφορά την χρήση των πόρων για τον έλεγχο, η δήλωση αξιοπιστίας καταναλώνει 50% περίπου των πόρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το Λεκτικό Συνέδριο για τη δήλωση αξιοπιστίας μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα μας όπου εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες για την μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Τώρα, όσον αφορά τον έλεγχο που κάνουμε για τις επιδόσεις. Πρώτα είπαμε ασχολιόμαστε με τη δήλωση αξιοπιστία. Στου ε, λοιπού πόρου του χρησιμοποιεί το ελεκτικό συνέδριο για να κάνει ελέγχου όσον αφορά τι ε, επιδόσει των διαφόρων οργανισμών. Είναι έλεγχοι οι οποίοι εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση σε διάφορου τομεί πολιτική και επικεντρωνόμαστε σε ιδιαίτερε πτυχέ ειδικού ενδιαφέροντο. Όπω είναι το κατά πόσο οι στόχοι που έχουν τεθεί έχουν επιτευχθεί όντω ή ποιο είναι το αποτέλεσμα διάφορων μέτρων που έχουμε υιοθετήσει. Επ' αυτού λοιπόν το ηλεκτρικό συνέδριο υιοθετεί πρόγραμμα για μια στρατηγική πολιετών ελέγχων που περιλαμβάνει διάφορους στόχους. Το... Η τρέχουσα στρατηγική μας, η πολιετές, υπάρχει αναλυμένη στην ιστοσελίδα μας. Κάνουμε λοιπόν τέτοιου ελέγχου επιδόσεων σε διάφορου τομεί, όπω σα είπα, όσον αφορά τι δαπάνε εκεί. Και κοιτάμε πώ καλύπτονται διάφοροι τομεί όσον αφορά του κινδύνου που ελοχεύουν. Για να προστατεύονται ακριβώ τα οικονομικά συμφέροντα των διαφερομένων. Επίσης, κοιτάμε να δούμε τι έχει γίνει και με την λήψη πολιτικών αποφάσεων και τους στόχους που έχουν επιτευχθεί από αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, Διάφορα θέματα που εξέτασε το Ελληνικό Συνέδριο για να δει κατά πόσο τα χρήματα πιάνουν τόπο είναι ε, διατροφική βοήθεια, επισητιστική βοήθεια μάλλον, για τους έχοντες ανάγκη, η διαχείριση της Επιτροπής ε, όσον αφορά προγράμματα Life και Nature, επίσης ενημέρωση και προώθηση ε, αγροτικών προϊόντων και διαχείριση τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποθήκευση δημητριακών. Εξετάσαμε επίσης την εφαρμογή των ποσοστών, των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων στα νέα Και στον τομέα της αλίας επίσης εξετάσαμε τον έλεγχο, την επιθεώρηση και τις κυρώσεις που επιβάλλονται όσον αφορά την διατήρηση των ειδών. Και τέλος υπάρχει και μια έκθεση που κάναμε πριν από δύο χρόνια περίπου ολοκληρώθηκε όσον αφορά την ε, ε, πολλαπλή συμμόρφωση, κατά πόσο είναι μια αποτελεσματική πολιτική ή όχι. Όλοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν οδηγήσει σε ειδικέ εκθέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, βρίσκονται και στην ιστοσελίδα μας. Επιπλέον, το ελεκτικό συνέδριο, και ίσως εδώ θα πρέπει αυτό να σας το πω πολύ σιγά, ότι πολύ σύντομα θα δημοσιεύσουμε ειδική έκθεση όσον αφορά το γαλακτοκομικό τομέα, την αγορά δηλαδή γαλακτοκομικών προϊόντων. Υπάρχουν ε, και άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε επιμονή μου βάσεως και θα ολοκληρωθούν ε, σύντομα, όπως είναι το πρόγραμμα LEADER, η ασφάλεια στον αφορά το κρέας, μέτρα συνδυασμένα γεωργία περιβάλλων, εκαθάριση ε, λογιστικών διαδικασιών, ίσπραξη πληρωμών που έχουν γίνει χωρίς να πρέπει και τέλος η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγοράς ζάχαρης. Το Ελεκτικό Συνέδριο ετοιμάζει το ετήσιο πρόγραμμά του για το 2010. Όταν θα έχει εγκριθεί από το Ελεκτικό Συνέδριο, το πρόγραμμα αυτό εργασία θα σα παρουσιαστεί από τον κύριο Καλδέρα, τον Πρόεδρό μα, κατά πάσα πιθανότητα τον Ιανουάριο του 2010. Τέλος, εκ μέρους του πρεσβύτερου της ε, ομάδας ελέγχου αριθμός 1, τον κύριο Γέσια Χάλας, θέλω να σας πω ότι εκφράζει την ε, θλίψη του που δεν μπόρεσε σήμερα να έρθει ο ίδιος αυτοπροσώπος να σας κάνει την παρουσίαση αυτή, αλλά υπόσχεται να έρθει κάποια άλλη στιγμή, εφόσον το επιθυμείτε. Εννοείται και τα άλλα μέλη της ε, ομάδας είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την προσοχή σας και ευχαρίστω να σας απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ελπίζω να μην ξεπέρασα το χρόνο που μου διαθέσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλεια, τέλεια. Τηρήσατε το χρονοδιάγραμμα τέλεια. σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσουμε, περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσης διάταξη, ζήτησε να παρέμβει Ο κύριο Χάσουερτ. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ το ελεκτικό συνέδριο και του ελεγκτέ για αυτά που κάνουν. Ξέρω, ασχολούνται με τη δήλωση αξιοπιστία κυρίω, σαν μέλο. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύτιμο να μάθω τα εξή. Ξέρω, Αναφέρθηκε για έλεγχο επιδόσεων και ποιότητα δαπανών, την αντιλαμβάνομαι εγώ. Θα ήταν καλό εμείς αμέλη αν ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις τους. Ποιότητα δαπανών, πώς χρησιμοποιούνται οι δαπάνες. Και θα βοηθούσε πολύ τα μέλη, πάρα πολύ, αν το ελεκτικό συνέδριο μπορούσε να δείξει ακριβώς ποιος κάνει τα λάθη. Στη Γεωργία δεν ισχύουν αυτά που λένε για τους πάντες. Αν μπορούσαν να κατονομάσουν θα μας βοηθούσαν πάρα πολύ, θα βοηθούσαν πάρα πολύ τη δουλειά που κάνουμε. Θέλετε κύριε Φένεση να απαντήσετε. Όχι, καλώς. Πολύ καλά. Πάμε λοιπόν πιο μπροστά και πάμε στο σημείο 6 της σημερινής διάταξης, διότι όπως σας είπα το θέμα για την ποιότητα θα το συζητήσουμε τελευταίο το σημείο 6 είναι ένα σημείο σημαντικότατο. Και αυτό προσέξτε το. Αφορά τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη, επικαιροποίηση ε, του οδικού χάρτη αν θέλετε. Το γάλα ήταν ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα. Ήδη εδώ και πολλά χρόνια οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έγιναν πολύ πτυτικές, ευμετάβλητες. Η συνεχής μείωση των αγροτικών τιμών που παρατηρήθηκαν κατά τελευταία 30 χρόνια διεκόπη το 2007 με μια αύξηση των τιμών που έφτασαν σε πολύ σημαίες τιμές τέλος 2007, αρχές 2008. Από τον Απρίλιο 2008 καταγράφεται για πολλά γεωργικά προϊόντα μια μείωση των τιμών τους. Όμως η διαθετική συγκυρία που ευνόησε την αύξηση των τιμών για τα γεωργικά προϊόντα φαίνεται να μπορεί να συνεχιστεί επί της βάσης μιας πρόβλεψης αυξήσεων ακόμα μεγαλύτερων που αναμένονται την επόμενη δεκαετία. Άρα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είδαμε στην περίπτωση του γάλακτος. Σήμερα θα πρέπει να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπασκιού. Μου λένε ότι ο κύριος Μπασκού καταφθάνει, έχει καθυστερήσει πέντε λεπτά. Όμως αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο, καλό, να σταθούμε στο θέμα της σπιτικότητας των τιμών. Ο κ. Μπασκού όταν φτάσει θα μας μιλήσει για τον οδικό χάρτη ή το, την ομάδα υψηλού επίπεδου για την ανταγωνιστικότητα του τομέα της παραγωγής των τροφίμων και μπορεί να μας δώσει σε αυτό το πλαίσιο κάποιες ενδείξεις. Όμως είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη το θέμα της μεταβολής των τιμών. Μπορώ να το κουβεντιάσουμε λίγο μέχρι να έρθει και ο Μπασκού. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε αρκετά, διότι βλέπουμε τι γίνεται με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και την αποσύνδεση. όλα αυτά οδήγησαν σε μια απτητικότητα των τιμών που δεν είχαμε συνηθίσει. Το βλέπουμε στο γάλα, ότι είχαμε κάποια θετικά μηνύματα, όπω μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν αυτά, αλλά αναφυσβήτητα αυτά τα θετικά μηνύματα καταφθάνουν αργά. Και οι παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να αντισταθούν πάντα όταν περνούν τι ε, δραματικέ στιγμέ των χαμηλών τιμών. Το θέμα του πώ να χειριστούμε την κίνδυνο στη Γεωργία, πώ να χειριστούμε το ευμετάβλητο των τιμών είναι κάτι που θα μα απασχολήσει σίγουρα. Α δώσουμε το λόγο στον κύριο Πασκού που έφτασε και μετά θα ακούσω τις δικές σας παρεμβάσεις. Θα σταματήσουμε για μερικά λεπτά. Γκαρσία, αν θέλετε να πάρετε το λόγο, κυρία. Ναι, Πρόεδρε. Αυτή η σύγκληση για το θέμα των τιμών στην Ευρώπη έχει να κάνει με την απόφαση και με αυτό που ζήτησε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας για το παρατηρητήριο των γεωργικών τιμών. Ο κύριος Βασκού θα μας μιλήσει για τη δημιουργία αυτού του παρατηρητηρίου τιμών, έτσι δεν είναι. Ελπίζω ναι. Θα τον ακούσουμε τώρα. Ελπίζω ναι. Εδώ έχουμε απλώς τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαν ένδειξη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα από πλευρά πολιτικής, διότι ασχοληθούμε σίγουρα με αυτό το θέμα στο μέλλον. Το πρόβλημα του πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτή το ευμετάβλητο των τιμών, πέραν από τις σωστές πληροφορίες, μέσω παρατηρίου κλπ. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει. Γι' αυτό ζητούσα να το προσέξετε. Να ξεκινήσετε τον προβληματισμό σας επ' αυτού. Ζητήσατε το λόγο. Είδα να σηκώνετε το χέρι σας. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ταιριάζει με αυτά που συζητούσαμε λίγο. Η της ισρών και Κροών. Μπαίνει χειμώνα. Και κτηνοτρόφοι χρειάζονται πρωτεΐνη. Και η πρωτεΐνη όλο γίνεται ακριβή, πιο ακριβή. Διότι ε, οφείλεται στη στάση των Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι της σόγιας και των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Τον περασμένο μήνα διώξανε τέσσερα καράβια ε, με σόγια γιατί είχαν γενετικά τροποποιημένα σόγια, είχαν ίχνη. Δεκάμιση εκατομμύρια λίρες κοστίζει κάθε φορά που γίνεται αυτό. Δεν θα στείλουν ξανά αυτά τα φορτία, οπότε ανεβαίνει η τιμή της σόγιας. Αν θέλετε να μειώσετε την πληθυκότητα, δείξτε κοινή λογική όσον αφορά το θέμα. Έφτασε ο κύριος Μπασκού και του δίνω με τα χαρά στο λόγο για να μπορέσει να συμμερώσει όσον αφορά τον οδικό χάρτη και μετά την παρέμβαση του κυρίου Μπασκού που έφτασε, λέει ο κ. Μπασκού, κατέφτασε. Και του δίνουμε το λόγο και μετά την παρέμβασή σας ε, θα, ακούσουμε την... θα ακολουθήσει η συζήτηση. Έχετε το λόγο, κύριε Μπασκού. Merci, Ζητώ συγγνώμη για αυτή την μικρή καθυστέρηση, αλλά είχαμε προβληματάκι συντονιστικό. Περιμένω να πάρει μπροστά υπολογιστή μου να βρω το password για να σας κάνω μια παρουσίαση του θέματος που είναι αρκετά τεχνικό. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την αναμονή εκείνης του υπολογιστού για να κάνω εισαγωγή στο θέμα. Θέμα της παρουσιάσεως είναι να σας δώσουμε μια εικόνα της πρόοδου που πετεύχει τον τομέα, της εφαρμογής του οδικού χάρτη, του roadmap. Είναι ένας οδικός χάρτης που κατατίστηκε και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2008 με σκοπό την ανάλυση, την εξέταση της λειτουργίας ε, του τομέα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτάθηκαν και κάποιες συστάσεις, έγιναν κάποιες πολιτικές προτάσεις που αποτελούν αντικείμενο του οδικού χάρτη. Πριν επισέλθω περισσότερο στο θέμα, να πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, ακόμα επεξεργαζόμαστε το θέμα της εφαρμογής του οδικού χάρτη. Δεν θα μπορούσα να σας παρουσιάσω λεπτομερώς όλα τα συμπεράσματα, τα πορίσματά μας και τις βασικές συστάσεις πολιτικής φύσεως που θα μπορούσαν να απορρεύσουν από αυτές τις εργασίες. Και το δεύτερο που έχω να πω ότι είναι επισέλθουμε στο θέμα, θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια πράγματα, να υπενθυμίσω κάπως το λόγο ύπαρξης του δικού χάρτη και από πού προέρχεται όλη αυτή η προβληματική του τομέα των τροφίμων. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή όλοι θα λάβατε αντίγραφο των διαφάνειών, θα βασιστώ στις διαφάνειες, θα θυμόσαστε ότι αν ξεκινήσαμε τη, εδώ και δύο χρόνια να επεξεργαζόμαστε πιο εντατικά τον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας είναι διότι το δεύτερο εξάμεινο του 2007 αντιμετωπίσαμε μεγάλη αύξηση των τιμών των γεωργικών προϊόντων και αυτό επέφερε πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών κατανάλωσης των τροφίμων και μετά τη μείωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων μετά το μέρος του 2008 είδαμε ότι ενώ είχαν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές κατανάλωσης των τροφίμων δεν μειώνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξήθηκε, στο ίδιο επίπεδο με τον οποίο αυξήθηκε και γι' αυτό εκφράζονται κάποιες ανησυχίες για τον τομέα, για τη λειτουργία. Τι γίνεται, πώς μεταβιβάζονται οι αλλαγές των τιμών μεταξύ παραγωγού, διανομέα μεταποιητού. Πώς γίνεται η κατανομή της προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα. Όχι μόνο μεταξύ γεωργού και διανομέων, αλλά μεγάλη διανομή και βιομηχανίας και μεταποίησης, αλλά υπάρχουν και ανησυχίε όσον αφορά τα διάφορα επίπεδα των τιμών που υπάρχουν στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα βλέπετε στην γραφική παράσταση διαφάνεια παριθμών 3 και στη διαφάνεια 4. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Εν συγκρίση με τη σημαντική αύξηση τη τιμή του γάλακτο τέλο 2007, τι τιμέ των βασικών προϊόντων, γαλακτοκομικών προϊόντων που μειώθηκαν κατά 50 με 60% σε ένα χρόνο. Ενώ οι τιμέ κατανάλωση των γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκαν μόλι κατά 1%. Είχαν αυξηθεί κατά 10% σε μερικού μήνε και εδώ και 1,5 χρόνο δεν αυξήθηκαν παρά μόνο κατά 1%. Δεν μειώθηκαν μάλλον κατά 1%. Άρα, τίθεται ερωτηματικό. Κατά πόσο λειτουργεί σωστά ο τομέας και στη διαφώνεια την επόμενη βλέπετε τη διαφορά τιμών που υπάρχει μεταξύ των βασικών προϊόντων στα διάφορα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές στις τάξεις του 60% όσον αφορά τις τιμές των τροφίμων, των απλών θα έλεγα, όπως είναι ο κοιμάς ε, του βοηίου, ε, χείριο κρέας, ψωμί. Άρα έχουμε ερωτήματα όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του τομέα και την αποτελεσματικότητα του τομέα. Και ξεκίνησαν κάποιες πρωτοβουλίες για αυτό το λόγο κατά τη διάρκεια 24-30 μηνών. Η πρώτη πρωτοβουλία ήταν η ανακοίνωση του Μαΐου 2008 που αφορούσε πιο συγκεκριμένα την παρακολούθηση του τομέα, την κερδοσκοπία, την εξέταση της λειτουργίας του τομέα. Ε, δεύτερη πρωτοβουλία που ξεκίνησε αφορά την ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2008 που πρότεινε τον περίφημο δικό χάρτη, το roadmap, με πέντε μεγάλες προτάσεις. Παράλληλα με αυτές τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγιναν κι άλλες. εργασίες του High Level Group for Food Competitiveness, ομάδα υψηλού επίπεδου, που επεξεργάστηκε το θέμα της ανταγωνιστικότητας του τομέα των τροφίμων, των γεωργικών προϊόντων και 2008-2009 συνεχίσαμε να εκμεταλλευόμαστε τις εργασίες που διεξήγονται όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σχετικά με τους μεγάλους διανομής. Υπήρξε σύγκληση των διαφόρων πρωτοβουλειών, κάτι που επέτρεψε φέτος να ρίξουμε φως όσον αφορά τη λειτουργία του τομέα αυτού για να επανέλθουμε στη διαφάνεια υπαριθμών 6, τον οδικό χάρτη, στον οδικό χάρτη είχαμε πέντε βασικές προτάσεις. Η πρώτη πρόταση είχε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του τροφίμων, των τροφίμων και της γεωργίας. Μετά να ενισχύσουμε την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε όλο τον τομέα. Τρίτη πρόταση. Εξέταση ενδελεχέστερη του ρυθμιστικού πλαισίου εντό του οποίου λειτουργεί ο τομέας στα διάφορα κράτη-μέλη. Τέταρτη πρόταση αφορούσε τη δημιουργία εργαλείου παρακολουθήσεως των γεωργικών και αγροτικοτροφημικών προϊόντων. Τρίτος, τρίτη πρόταση, να εξετάσουμε αν υπήρχε ανάγκη να θεσπίσουμε μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών της κερδοσκοπίας επί των ε, προϊόντων. Εργαστήκαμε πολλά όσον αφορά την ε, σύνταξη αυτών των πέντε προτάσεων. Θα ήθελα να αναφερθώ εκ νέου σε κάποιες από τις προτάσεις. Η πρώτη πρόταση αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα του αγροτροφημικού. Αυτή η πρόταση πάνω απ' όλα εφαρμόστηκε μέσω της ομάδας υψηλού επίπεδου High Level Group on Food Competitiveness που υιοθέτησε 30 συστάσεις, ένα σύνολο 30 συστάσεων, που θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες, τα δύο-τρία επόμενα χρόνια. Και αυτές οι προτάσεις, αυτές οι συστάσεις αφορούν πέντε βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα η αγροτική, περιβαλλοντική πολιτική. Δεύτερο θέμα η νέα αγορά και η λειτουργία της ενιαίας αγοράς στα πλαίσια των, στον τομέα των τροφίμων. Τρίτη πρόταση, λειτουργία του τομέα των τροφίμων, της βιομηχανίας των τροφίμων τέταρτη ομάδα συστάσεων ασχολείται με θέματα έρευνας και ενοτομίας. Πέμπτον, εμπορική πολιτική, εξαγωγές. Επεσεργαστήκαμε και τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων στο φορέα, στον τομέα. Έγιναν ακροάσεις με τους εμπλεκομένους στον τομέα, με τους ενδιαφερομένους και με το δίκτυο των αρχών ανταγωνισμού των διαφόρων κρατών μελών και επελήφθημεν διαφόρων θεμάτων. Πρώτα απ' όλα, της ύπαρξης πρακτικών αντιαντιαγωνιστικών σε κάποιους τομείς, σε κάποιες χώρες. Επεξεργαστήκαμε επίσης τις σχέσεις μεταξύ δυνατότητας διαπραγμάτευσης και πρακτικών αδίκων από την άλλη όσον αφορά τις εμπορικές πρακτικές που θα μπορούσαν να είναι άδικες έναντι κάποιων. Έγιναν κάποιες προσπάθειες λοιπόν και πιθανότατα θα καταλήξουμε σε συστάσεις που θα υποβληθούν τις επόμενες εβδομάδες. Τέταρτος τομέας εργασιών. Διαφάνεια. Να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο εποπτείας των τιμών δηλαδή. Όσα σχετίζονται με τη διαφάνεια λειτουργίας των παραγόγων προϊόντων δημιουργούμε εργαλείο παρακολούθηση των, τιμών σε όλο το τομέα, σε όλα τα κράτη-μέλη, κάτι που γίνεται εξάλλου σε κάποιες χώρες. Και κάναμε διάφορες προσπάθειες αναλυτικές όσον αφορά την κατανομή της προστιθέμενης αξίας σε όλη την αλυσίδα και τη διαφάνεια όσον αφορά τις τιμές. Είναι αρκετά τεχνικά θέματα θα παρουσιάσω τα βασικά συμπεράσματα των ε, αναλυτικών προσπαθειών. Εδώ και 15 χρόνια αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει αρκετά σημαντική μείωση του ποσοστού της γεωργίας όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της αλυσίδας. Πριν είχαμε 95% γεωργία στην προστιθέμενη αξία που παράγεται από τα αγροτροφομικά ε, προϊόντα και το 2005 ε, έπεσε κατά 24% διότι ο γεωργικός τομέας δεν μπόρεσε να εισπράξει από την αύξηση των τιμών. Οι ονομαστικές αξίες μείνανε σταθερές βέβαια επί περίπου 15 χρόνια. Άλλο συμπέρασμα για τη διαβίβαση, για τη μετακίνηση των τιμών. Επί 15 χρόνια δεν υπάρχει συσχετισμό μεταξύ του αγροτικού τομέα και βιομηχανία όσον αφορά τι τιμέ και του μεγάλου διανομή. Είναι αδύναμη η μετακύληση του κέρδου. Μικρή. Στα νέα κράτη-μέλη είναι πιο σημαντικό το φαινόμενο από ό,τι στα παλιά. Και βλέπουμε ότι αυτή η μετακύληση του κέρδου άλλαξε από φύση και εύρος, σε φύση και εύρος από το 2007 και μετά, μετά τη μεγάλη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών διότι βλέπουμε ότι έχουμε ένα, ένα φαινόμενο σύμφωνα το οποίο αυξήθηκαν τιμές των τροφίμων μετά την τιμή των γεωργικών προϊόντων το 2007, αλλά μετά το 2008, αρχές του 2008, είδαμε ότι οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν πολύ λίγο. Πολύ μικρή μείωση. Παρά τη μεγάλη πτώση των πρώτων υλών των γεωργικών υπάρχει πρόβλημα ασυμμετρίας, πρόβλημα ε, μετακύληση των τιμών στον τομέα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολο να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα που αναφορούν όλες τις χώρες και όλο τον τομέα. Κάθε αλυσίδα, κάθε ε, τομέας ανάλογα με το προϊόν και ανάλογα με τη χώρα έχει ιδιαιτερότητες. Και αυτή με ο αντίκτυπος που έχουν τιμές είναι πολύ μικρός και καμιά φορά δεν αντικατοπτρίζεται σε προβλήματα λειτουργία του τομέα, ίσως να οφείλεται σε κάτι άλλο. Στατικές των επιχειρήσεων, που λόγω μακροπρόθεσμων συμβάσεων που συνάπτονται, ακολουθούν αυτή την προσέγγιση. Διάφορα στοιχεία που οδηγούν σε κακή λειτουργία του τομέα και σε μικρή αποδοτικότητα. Άλλο σχόλιο. Όλες αυτές οι προσπάθειες σχεδόν τελειώνουν θα υποβάλουμε τις επόμενες εβδομάδες πιθανότατα έκθεση που θα αφορά τη λειτουργία του τομέα και θα δώσουμε πολιτικές συστάσεις. Θα υιοθετηθεί αυτό το έγγραφο μέχρι το τέλος του έτους 2009 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, κύριε Μπασκιού. Τον ευχαριστώ τον κύριο Μπασκιού για την παρουσίασή του αυτή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβαθύνουμε σε αυτή την ανάλυση που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι όπως βλέπουμε και στο γάλα και σε άλλους τομείς, πολλούς τομείς, έχουμε δραματική πτώση των τιμών των γεωργικών προϊόντων που δεν αντικατοπτρίζεται σε μια μείωση των τιμών κατανάλωσης. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που πολύ συχνά απασχολούν αυτή την Επιτροπή. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε στους λόγους για τους οποίους δεν καταφέρνουμε να, να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας σε αγροτικό επίπεδο. Ίσως είναι πτυχή αγροτική που αφορά τη δυσκολία να διοργανωθεί ο αγροτικός κόσμος από πλευράς συμβασιακής κλπ. Αλλά πρέπει να δούμε και στα διάφορα δίκτυα τα γεωργικά πού μπορούμε να εντοπίσουμε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η μεταφορά της αξίας, μετακύληση της αξίας ε, οδηγεί στους παραγωγούς και στους καταναλωτές, δεν δικαιολογεί να είναι αδύναμη μικρή και οι καταναλωτές και οι παραγωγοί. Θα ανοίξουμε τη συζήτησή μας, αλλά καλό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα εξετάσει βάθος αυτά. Διότι έχω την εντύπωση ότι το θέμα της πτητικότητας των τιμών θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Τώρα πλέον βλέπουμε διακυμάνσεις πολύ μεγάλες που δεν είχαμε συνηθίσει. Αλλά αν κάνουμε ένα χρονικό βήμα προς τα πίσω, πριν ξεκινήσει η κοινή αγροτική πολιτική δεκαετία του 60, ακριβώς αυτό συνέβαινε στις ευρωπαϊκές αγορές τότε. Η κοινή αγροτική πολιτική εισήχθη ακριβώς για να σταθεροποιήσουμε τις τιμές και τα εισοδήματα. Σήμερα με μια κοινή αγροτική πολιτική αποσύνδεσης και ενισχύσεως των εισοδημάτων επιστρέφουμε ξανά σε μια πολύ μεγάλη τέτοια διακύμανση. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά για να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε διαχείριση των κινδύνων για τους γεωργούς. Στάρντι, ο πρώτος αγορήτης. Ξεκινάμε τη συζήτηση. No, okay. Uh, thank you, uh, Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως πάντοτε δηλώνω το ιδιαίτερο συμφέρον που έχω, διότι μπορεί να είναι και δημοσιογράφοι εδώ. Είμαι γεωργός ε, είμαι και αναμειγμένο στην μεταποίηση και είμαι 15 χρόνια ευρωβουλευτής και μέλο τη παρούσης επιτροπή. Κύριε Μπασκή, διαρωτώ με, σε, σε ποιον πλανήτη ζείτε, μήπως δεν είστε στην γη. Οι εκμεταλλεύσει που γνωρίζω είναι business, δεν είναι για απόλαυση. Λέτε ότι έχουν σταθεροποιηθεί ή και μειωθεί τα κόστη της εκμετάλλευσης. Ίσως εδώ να υπήρξε κάποιο σφάλμα μεταφράσεως, αλλά σας υπενθυμίζω ότι η τιμή του πετρελαίου συνεχίζει να αυξάνεται. Άρα συνεχισει να αυξανεται αρα καυσιμα και ε, λιπάσματα αυξάνουν. Και εσείς έχετε ε, υιοθετήσει μέτρα τα οποία έχουν δραματικά αποτελέσματα στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί Πίτερ Μάντελσον οι γεωργοί εξασφαλίζουν το εισόδημά τους από την αγορά τηρώντας ακριβώς τα προβλεπόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τον γύρο του Ντόχα. Αλλά να σας εξηγήσω κάτι αν δεν το έχετε κατανοήσει. Ότι η γεωργία δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμείνει οικογενειακή εκμετάλλευση. Πρέπει να βγάλει λεφτά. Υπάρχουν έξοδα για τα μηχανήματα, για τα εργατικά χέρια και μόλις Τώρα ψηφίστηκε σημαντική νομοθεσία ευρύτατη εφαρμογή για τα λοιπάσματα που θα έχει βαρύτατε συνέπειε στι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Οι δικοί μου γεωργοί δεν θα συνεχίσουν να παράγουν τρόφιμα εάν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Θα το γυρίσουν στην παραγωγή ενέργεια. Έχετε λοιπόν κοιτάξει εσεί η Επιτροπή την ασφάλεια των τροφίμων. Μέχρι πότε θα παράγουμε φθηνά. Ο ε, πρόεδρος είπε και σωστά ότι δεν έχει επωφεληθεί ο καταναλωτής από την μείωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Θα είναι παγκόσμιες οι τιμές των γεωργικών προϊόντων. Ακόμα και εάν κάτι το πουλάμε 100 ε, ευρώ τον ε, τόνο, το 2007 είχαμε τα διπλάσια το αποτέλεσμα ήταν διπλέσια τιμή. Και μιλώ για το σιτάρι. Η, τιμή του ψωμιού μας δεν αυξήθηκε. Η γεωργία λοιπόν θέλει να εξασφαλίσει τα προστοζήνη και αυτό πρέπει να το κάνει από την αγορά. Άρα πρώτα πρέπει να εξασφαλίσετε την ασφάλεια προμήθειας τροφίμων και ακόμα πιο σημαντικό να εξασφαλίσετε ώστε οι γεωργοί να μπορούν πραγματικά να εξασφαλίσουν τα προστοζήν από την αγορά. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι εμένα με απογοήτευσε κάπως όλο αυτό που μας είπε ο υπάλληλο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί ήδη πριν από τις εκλογές, πάνω από 7,5 χρόνια είμαι εδώ βουλευτής αυτή την Επιτροπή, πολλές φορές λοιπόν έχω ακούσει τα ίδια συμπεράσματα όπως αυτά που σήμερα μας, μεταφέρατε εσείς. Ε, εμείς θέλαμε να ξέρουμε αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις τιμές της αγοράς και εκείνες που παίρνουν οι παραγωγοί. Γι' αυτό και κάναμε η κυρία Μπατζελή που ήταν η μία, και εγώ συνεργάστηκα μαζί της, έκθεση πρωτοβουλίας λοιπόν, και σε αυτήν την πολύ ωραία έκθεση πρωτοβουλίας που με τεράστια πλειοψηφία εγκρίναμε, ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα παρατηρητήριο τιμών είναι κάτι που πολύ εύκολα μπορείτε να κάνετε με τα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας και έτσι θα μπορούσαν οι παραγωγοί να καταδείξουν κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι χρειάζεται να καταπολεμηθούν οι παράτυπες ε, διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα. Γιατί αυτά που μας είπατε εσείς ότι από 31 πήγε 24% το κομμάτι που παίρνει ο παραγωγός Μα δεν είναι ότι θέλουν ε, αύξηση των τιμών οι αγρότες, δεν είναι αυτό που θέλουν, εξάλλου υπάρχει και διανομή που δεν τους το επιτρέπει. Αλλά να, εδώ θα το θυμόσαστε κι εσείς, σε άλλη έκθεση που κάναμε είδαμε, σε μία κρόαση μάλιστα επίσης εδώ, πώς φτάνουν σε αυτή την κατάσταση οι αγρότες. Χρειαζόμαστε ελεύθερο ανταγωνισμό και ακριβώς επειδή χρειαζόμαστε και κοινωνική οικονομία και στη Γεωργία, γι' αυτό η παραγωγή ζητούν ξανά και ξανά την δημοσίευση των αγροτικών τιμών. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε είναι να έχουμε αυτό το παρατηρητήριο τιμών. Πρέπει να το φτιάξετε. Αν δεν το κάνετε από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο, όπου θα πρέπει να αποφασίσει το Κοινοβούλιο, θα πρέπει ξανά να κάνουμε έκθεση πρωτοβουλίας για να σας ξαναπούμε ότι πρέπει να ακούτε τη φωνή των πολιτών, των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να φροντίσουμε να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε. Ευχαριστούμε. Άλμπερντες. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τυχαίνει να έχω εδώ μπροστά μου ορισμένε στατιστικές, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε, Βέβαια αναφέρονται στη Γερμανία και σίγουρα δεν αφορούν όλες τις χώρες μέλη τη Ένωση και πάντω όχι τις νεότερες. Ωστόσο Πρόκειται για μια σύγκριση μεταξύ 1970 και 2007. Και όπως ελέγχθη ήδη πριν, το 1970 στην Γεωργία είχαμε συμμετοχή των γεωργικών προϊόντων στη, στη, στην, ε, στη ζήτηση του καταναλωτού 47% το 2007 έχει πέσει. Σημαντική είναι και η στατιστική για τις τιμές των, ε, του ΣΥΤΟΥ. Το 2008 είχαμε σχετικά καλές τιμές για τα στάρια. στατιστική είναι ως εξής. Το 1970 ένα κιλό δημητριακά ήταν 18 σέντ. Ακριβώς την ίδια τιμή όπως το 2007 όπου ήταν πάλι 18 σέντ, 18 λεπτά. Η τιμή όμως του καταναλωτού έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το 1970 ήταν 66 σέντ, 66 λεπτά το 2007 είναι 250 για τον καταναλωτή. Δηλαδή σχεδόν 300% παρόλο που η τιμή του σταριού παρέμεινε ακριβώς ίδια. Η τιμή του ψωμιού όμως αυξήθηκε. Τι μας λέει αυτό. Σημαίνει ότι αυτά που λαμβάνει τελικά ο Γεωργός έχουν πολύ, η τιμή του Γεωργού δηλαδή, έχει πολύ, χαμηλή, πολύ μικρή συμμετοχή στην τιμή του καταναλωτού. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να αυξηθεί το μερίδιο από την τιμή αυτή του γεωργού χωρίς να υποστεί ζημιά ο καταναλωτής. Το σημαντικό είναι, το ενδιαφέρον είναι ότι στη Γερμανία για έναν μέσο εργάτη της βιομηχανίας τα τρόφιμα έχουν φτηνίνει σημαντικά. Έχω εδώ πάλι στατιστική, 8 τρόφιμα με όλες τις λεπτομέρειες, εγώ δεν θα τις πω τώρα, αλλά πρόκειται για το ίδιο καλάθι τροφίμων το 1971 ένας εργάτης βιομηχανίας έπρεπε να δουλέψει 4 ώρες και 3 λεπτά και το 2007 1 ώρα και 15 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές στην Γερμανία χρειάζεται να ξοδέψουν αναλογικά όλο και λιγότερα από ε, το εισόδημά τους για, για την διατροφή τους. Έχουμε φτάσει σήμερα στο 11%. Άρα οι καταναλωτές ασφαλώς και έχουν υποφεληθεί από την εξέλιξη αυτή. Και γι' αυτό και άλλωστε είναι δικό μας καθήκον αυτό να φροντίσουμε ώστε και η γεωργία να λάβει το μερίδιο που της αξίζει από την εξέλιξη αυτή έτσι ώστε στο μέλλον να συνεχίσουν να μπορούν να υπάρχουν και να λειτουργούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ Άλμπερτ. Γεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους γεωργούς μας, αλλά και για μας, διότι εδώ διακυβεύεται η αξιοπιστία των πολιτικών. Εμείς θέλουμε να υπάρξει η γεωργία. Θέλουμε να μπορεί να λειτουργήσει και μέσα στην οικονομία της αγοράς. Θέλουμε οι γεωργοί να μπορέσουν να κατακτήσουν τις αγορές τους. Και βεβαίως έχουν ε, την αξίωση να τους δίνονται αξιοπρεπείς τιμές. Από την μια μεριά μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, και επομένω οι γεωργοί πρέπει να αναζητήσουν άλλε πηγές εισοδημάτων. Αυτό είναι και το αποτελεσματικότερο μέτρο, να μπορεί ο ίδιος ο Γεωργό να αποφασίσει εάν θα πουλήσει τα δημητριακά του στον έμπορο δημητριακών ή εάν θα ε, τα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή ενέργεια. Αυτό ε, θα το καταλάβει. Διότι τότε και ο Γεωργός θα πουλήσει το δημητριακό του στον έμπορο μόνο αν αυτός προσφέρει καλύτερη τιμή. Τώρα, όταν οι διακειμενόμενες τιμές και εφόσον δεν ε, υπάρξει μετακύληση της τιμής εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι απάτη θα πρέπει να υπάρχει κάποια διασύνδεση και εφόσον υπάρχουν, υπάρχει αύξηση των τιμών καταναλωτού θα πρέπει αυτή να έχει μια πύχηση και στην τιμή του Γεωργού τι μπορούμε να κάνουμε νομίζω ότι το καλύτερο όπως είπε και η συναδελφός μου εδώ η κυρία Γκασία είναι είναι να ανοιχτούν τα χαρτιά, να ε, γίνει ανοιχτή συζήτηση. Να μιλήσουμε ανοιχτά και καθαρά. Διότι αυτό θα κατανοήσουν όλοι. Οι δεμοί, όσοι δεν τα καταφέρουν, θα παραμείνουν στην άκρη του δρόμου. Εγώ έχω και ένα άλλο ε, παράδειγμα που λέω συχνά σε συναντήσεις γεωργών. Εάν διπλασιαστεί η τιμή του Δημητριακού εν τέλει η τιμή του Γιώργου θα αυξηθεί κατά 1%. Η τιμή του Κανατολτού θα αυξηθεί κατά 1%. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει διαρκώς η εντύπωση και δικαιολογημένα ότι ε, γίνεται εκμετάλλευση σε βάρος του Γιώργου. Ζωζέ Μποβέζη, το λόγο. Ζωζέ πρώτα και μετά κυρία Πόλσον. Ναι, εκπλήσωμε εκπλήσωμαι από αυτά που υπόθηκαν όσον αφορά τις τιμές και τα εργαλεία για να υπάρξει μια κάποια τοποθέτηση των πραγμάτων στη θέση τους. Να πω ότι ε, οι παγκόσμιες τιμές ποτέ δεν ήταν οικονομικές τιμές. Οι τιμές σε παγκόσμια αγορά ήταν τιμές πολιτικές, dumping. Το βλέπουμε στο γάλα, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα όσον αφορά τη Νέα Ζηλανδία. 1% της παραγωγής καταστρέφονται οι τιμές. Σήμερα το πρόβλημα της Ευρώπης ποιο είναι. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ δεχτήκαμε οι εσωτερικές τιμές να είναι οι τιμές της αγοράς, της παγκόσμιας αγοράς. Ξεκινώντας από εκεί, είμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να φτιάξουμε μια πραγματικότητα τέτοια ε, όσον αφορά τι τιμέ, το επιτρέπει στου γεωργού να καλύψουν το κόστο παραγωγή. Έχω την εντύπωση ότι όπω τίθεται η συζήτηση, κυρίω αυτό το έγγραφο, είναι για την αγροβιομηχανία αυτό το έγγραφο και όχι για τους αγρότες. Αν συνεχιστεί η διαδικασία στην οποία έχουμε μπει και αύριο θα έχουμε παγκόσμια προμήθεια προϊόντων στον κόσμο, αλλά δεν θα έχουμε κανένα γεωργό στην Ευρώπη. Δεν είναι αγροτική πολιτική αυτή, αλλά είναι πολιτική που ακολουθούμε προ όφελο του αγροτροφημικού τομέα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε στις βασικές μας αρχές. Ευχαριστώ, Ζώζε. Η κυρία Πόλσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι γεωργοί στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο αντιμετωπίζουν μάλλον απαρτίζονται από πολύ μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων, μικρών εκμεταλλεύσεων. Και αυτοί που εισακούγονται είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Οι πολύ μεγάλες βιομηχανίες παγκοσμίου εμβέλειας που έχουν τα μέσα να παράγουν χημικά προϊόντα, λιπάσματα κλπ. Τεράστιες επιχειρήσεις είναι αυτές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και η γεωργία τελικά δεν είναι τόσο σημαντική. Η γεωργία λοιπόν προσπαθούν να συνενωθούν, να φτιάξουν επιχειρήσεις. Η γαλακτοπαραγωγή πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά είναι έρμεα στα χέρια της Πάρμα, ΛΑΤ και άλλων παρομοίων εταιριών. Και φαίνεται να αποκτούν όλο και μικρότερη σημασία. Θα πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε γιατί οι γεωργοί γιατί οι γεωργοί, λέγω, βρίσκονται σε μια τέτοια θέση όσον αφορά την παραγωγή τροφίμων. Ο ανταγωνισμός δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα από μόνος του. Έχουμε μια λυσίδα ενδιαμέσων που παρεμβάλλονται μεταξύ γεωργού και καταναλωτού. Νομίζω λοιπόν ότι ίσως δεν πρέπει να απορριθμίσουμε την ε, γεωργία, το τομέα της γεωργίας, αλλά να τον ρυθμίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι τώρα δεν μπορούμε να απαιτούμε να επανέλθουμε στο παρελθόν καθεστώς. Δεν μπορεί να ισχύσει αυτό που είχαμε στο παρελθόν στο μέλλον, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε μηχανισμούς σταθεροποίησης των τιμών. που οι τιμές ποικίλουν απρόβλεπτα. Κυμαίνονται απρόβλεπτα. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν μέτρα που θα υπερασπίζονται τον τομέα και θα σταθεροποιούν την αγορά προς όφελος των γεωργών, οι οποίοι οι γεωργοί υποφέρουν. Υποφέρουν από την πτώση των τιμών. Ίσως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο ασφαλείας ασφαλίσεων όπως έχουμε για τις καταστροφές, την ξηρασία, τις πλημμύρες κλπ. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε ε, υπό συνθήκες, με νέους όρους, να εξετάσουμε το θέμα. Ευχαριστώ κυρία Πόλσεν. Πολύ σημαντικό να σκεφτούμε νέα μέσα, νέα εργαλεία, διότι το θέμα τη διακύμανση των τιμών θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με νέα μέσα, όχι του παρελθόντος. Κανείς δεν θέλει να επιστρέψουμε στα μέσα του παρελθόντος, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε νέα μέτρα, τα οποία θα μπορέσουν να σταθεροποιήσουν το εισόδημα των γεωργών και την παρέμβαση, με μια προσέγγιση που θα είναι πιο κοντά στη γεωργία. Σμιτ, ο κύριος Σμιτ έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Ζωζέ και ο Ρόμπερτ Στέρντι. Εγώ βέβαια θα τα πω λίγο πιο ευγενικά στον εκπρόσωπο της Κομισιόν από ότι ο Στέρντι. Υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στην κοινή αγροτική πολιτική και στις τιμές της αγοράς. Είναι σαφές και το Κοινοβούλιο το έχει ξεκαθαρίσει αυτό και είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται να το μελετήσουμε. Ασφαλώς και γίνονται προσπάθειες έγραψα μια φράση που είπατε, ότι δεν μπορεί κανείς να συναγάγει συγκεκριμένα συμπεράσματα, διότι υπάρχουν ιδιωτερότητε των διαφόρων αγορών. Ναι, υπάρχουν βέβαια, αλλά οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούμε είναι κοινοί για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο τρόπος με τον οποίο εκπροσωπεί, για παράδειγμα στον ΠΟΕ, η, ε, η Κομισιόν την κοινή αγροτική πολιτική, είναι ακόμα πιο κοινό. Υποτίθεται ότι έχουμε ένα οδικό χάρτη και αυτό ο οδικό χάρτη υποτίθεται ότι πρέπει να έχει ένα προορισμό. Εγώ δεν βλέπω προορισμό στι διαβουλεύσει που έχουν γίνει μέχρι τώρα. σω αυτά να εκπονούνται ακόμα και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Αλλά με ανησυχεί κάπω. Ότι δηλαδή ενδέχεται απλώ να γίνει άλλη μια μελέτη που δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πρόκειται να γίνει θεμελιώδη αναδιάρθρωση τη ε, κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε ακούσει, ακούσει ήδη για του διάφορου ε, στόχου που μελετάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εγώ νομίζω ότι έρχονται σε αντίθεση με την ασφάλεια τροφίμων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που αυτό με απασχολεί διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν α, συνεννοούνται. Και εν τέλει αυτοί που χάνουν είναι η παραγωγή. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Θα είναι έτοιμα αυτά μέχρι τέλους του έτους και θα περάσουν στις μελλοντικές συζητήσεις για το πού θα πάει η κοινή αγροτική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρήσει ότι πρόκειται για σημαντική προτεραιότητα μέσα στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, ότι πρέπει το κενό αυτό, η απόσταση αυτή ανάμεσα στις τιμές της ε, ε ΚΑΠ και της αγοράς θα αντιμετωπιστούν ή θα δούμε εν τέλει 20 διαφορετικές προτεραιότητες να προτείνεται, οι οποίες δεν θα συμμορφούνται μεταξύ τους. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Κλείνουμε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Βοητσοβόσκη, τον κύριο Αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Είναι καλό που έγινε αυτή η συζήτηση σήμερα και νομίζω ότι σταδιακά ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει ανάγκη να γίνει μια συζήτηση αρχών για την Γεωργία. Είμαι για δεύτερη θητεία Ευρωβουλευτής και οφείλω να πω ότι τα προηγούμενα πέντε χρόνια τα περάσαμε συζητώντας μεταρρυθμίσεις που οδηγούν εν τέλει στην σταδιακή κατάργηση της γεωργίας. Δεν πρόκειται για την, αγορά, για την οργάνωση αγοράς του κρασιού ή της ζάχαρης. Αυτό που μας απασχολούσε κυρίως ήταν η μείωση της παραγωγής. Πώς θα πείσουμε τους γεωργούς να μειώνουν την ε, παραγωγή. Στο μεταξύ, οι εταίροι μας κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Εγώ μετέβην στην Ιαπωνία και είδα να ε, καλλιεργούν ρύζι και στο τελευταίο τετραγωνικό ελεύθερο μέτρο. Ακόμα και στα σπίτια τους φυτεύουν ρύζι. Υποτίθεται ότι είναι χαμηλέ τιμέ του ρυζιού. Ε, μα τότε γιατί το κάνουν. Και γιατί δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα εδώ στην Ευρώπη. Εγώ ρώτησα τους γεωργούς Τρία αμερικανικά δολάρια το κιλό το ρύζι. Πιθανώς η τιμή αγοράς του ρυζιού είναι υψηλότερη από ότι η τιμή του τελικού καταναλωτή. Ναι, ερχόμαστε όμως τότε στο ίδιο βασικό ερώτημα. Θέλουμε να έχουμε γεωργία ή όχι. Διότι στην πραγματικότητα συμπεριφερόμαστε σαν δήθεν να ενδιαφερόμαστε για την γεωργία. Στην πραγματικότητα όμως οι προσπάθειες που κάνουμε εδώ από κοινού είναι η μείωση, η κατάργηση εν τέλει της γεωργίας. Κανείς δεν συμφωνεί να διαλυθεί αυτή η Επιτροπή, αυτό θα επεξεργαστούμε, αυτό θα... αυτή η προσπάθεια θα κάνουμε. Θα δώσω για κάποια λεπτά το λόγο στον κύριο Μπασκού για να δώσει μια σύντομη απάντηση και μετά πάμε στο επόμενο σημείο της σας διάταξης. Κύριε Μπασκού, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις και για τις προτάσεις που κάνετε. Θέλω να απαντήσω σε δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ναι, προβλέπετε και γι' αυτό και λυπάμαι που τη συζήτηση την κάνουμε τώρα, γιατί είμαστε στο τελικό στάδιο προετοιμασίας των ε, ερευνών αυτών και των πολιτικών συστάσεων που μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου θα κοινοποιηθούν. Αν δηλαδή είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση σε έναν άμιση μήνα, θα είχα περισσότερα στοιχεία να σας δώσω πιο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα για το παρατήριο τιμών στο οποίο αναφερθήκατε πολλοί από εσά. Πράγματι μέχρι τα τέλη της χρονιάς κάτι θα έχουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και θα τα δούμε μέσα στους επόμενους μήνες. Πάντως, το θέμα αυτό που έχει να κάνει και με τα τρόφιμα είναι θέμα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σπάνια έχω δουλέψει τόσο πολύ και συνεργαστεί με τις άλλες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμός, Εσωτερική Αγορά, Πολιτική Καταναλωτών, Στατιστική Υπηρεσία, ε, Οικονομικά και Χρηματοπιστωτικά Ζητήματα. Πραγματικά η δουλειά που έχει γίνει, έχει γίνει σε βάθος. Φυσικά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μας, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας παρουσιάσω κάτι συγκεκριμένο. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ότι όλοι ζούμε στον ίδιο πλανήτη, όμως δεν μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα και νομίζω ότι διαφορετικά καταλαβαίνουμε την παραγωγή. Άλλοι λένε ότι μειώθηκε, μα όντως εδώ και αρκετό καιρό γίνεται αυτό, αλλά η αγορά αντικατοπτρίζει αύξηση με τις τιμές που έχουν αυξηθεί. Θέλω εδώ να σας πω ότι το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής στην τελική τιμή μειώνεται. Αυτό βέβαια είναι ένα μηχανικό φαινόμενο. Το υπόλοιπο κόστος, ενέργεια, εργατικό δυναμικό, κεφάλαιο, το κόστος αυτό αυξάνει συνεχώς. Οπότε, δεδομένου ότι δεν αυξάνονται οι αγροτικές τιμές ιδιαίτερα, καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι του γεωργικού προϊόντος στο τελικό, στην τελική τιμή, μειώνεται. Εξάλλου, όλο και περισσότερο καταναλώνουν μεταπημένα προϊόντα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Οπότε, ο γεωργικός τομέας ε, κερδίζει λιγότερο. Τέλος, είναι θέμα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το ζήτημα. Θα προτείνουμε σύνολο πολιτικών συστάσεων που θα βασίζονται στις έρευνες που κάνουμε, στις μελέτες που κάνουμε. Αλλιώ οι αποφάσεις δεν θα είναι καλές. Όλα αυτά θα τα έχουμε τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Καλώς. Ελπίζουμε πολύ γρήγορα να έχουμε ε, νέα μαντάτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε λοιπόν στο σημείο 5. Ή μάλλον να επιστρέψουμε στο σημείο 5, διότι ο κύριο Τζανκάρλο Σκότα εν τω μεταξύ κατέφθασε. Θα μιλήσουμε για την ποιοτική πολιτική, πολιτική ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η έκθεση είναι μια απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις πολιτικές για την ποιότητα που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που προτάθηκαν το 2009. Εγώ τι θα έλεγα να κάνουμε, να δώσω το λόγο αμέσως στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην κυρία Μπενίτε Σάλας της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργίας και μετά θα περάσουμε στον κύριο Σκότα, ο οποίος θα μπορέσει να μας παρουσιάσει την έκθεσή του και εν συνεχεία ξεκινάει η συζήτησή μας. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Μπενίτες Σάλας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Πολύ σύντομα. Θα συνοψίσουμε την πολιτική ποιότητα γεωργικών προϊόντων που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που μας ζητήσατε είναι μια τεχνική παρουσίαση ώστε να εξοικειωθείτε περισσότερο με τα θέματα επικαιρότητα που εξετάζεται ήδη. Θα ξεκινήσω λοιπόν πρώτα απ' όλα υπενθυμίζοντας λιγάκι πώς έχει προχωρήσει η πολιτική μας αυτή. Τη δεκαετία του 60 και του 70, όπου και αναπτύχθηκαν οι πρώτες προδιαγραφές ε, τυποποίησης με τις ε, κοινέ οργανώσεις αργοράς και στη συνέχεια τη δεκαετία του 80 που είχαμε τις πρώτες προδιαγραφές για τις ετικέτες των προϊόντων, ώστε να έχουμε ποιότητα ιδίως το κρασί. Και μετά είχαμε τη δεκαετία του 90 όπου είχαμε επίσης προδιαγραφές ποιότητας, εθελοντική βάση, βιολογική παραγωγή, παραγωγή ποιότητας και την περίφημη ονομασία προελεύσεως για προστατευμένα προϊόντα στην αγορά μας. Στη συνέχεια είχαμε διάφορες κρίσεις ε, που είχαν να κάνουν με την υγεία του καταναλωτή, οπότε ασχοληθήκαμε περισσότερο με την ασφάλεια των προϊόντων και μετά από τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής είχαμε και το περίφημο θέμα της πολλαπλής συμμόρφωσης που οδήγησε στις ρυθμίσεις υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και υπέρ της ποιότητας των προϊόντων. Έτσι λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 90 ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο ομάδες κανόνων η μία ομάδα υποχρεωτική που αποτελεί το κοινό βάθρο, ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, με την υγιεινή των ζώων και το περιβάλλον και μετά έχουμε και ορισμένα μέσα σε θελοντική βάση που είναι η ονομασία προέλευσης, η γεωγραφική προέλευση κλπ. Το καθένα έχει και το δικό του λογότυπο για να γίνεται πιο εύκολα διαφοροποίηση στην αγορά. Τώρα η ανάπτυξη αυτή με τα χρόνια οδήγησε βέβαια σε πολυπλοκότητα της πολιτικής μας. Γιατί οι προδιαγραφές εμπορίας αναπτύχθηκαν σιγά σιγά όλα αυτά τα χρόνια και αυτό έγινε όμως κατακαιρματισμένα, ανατομέα και όχι καλά συνδυασμένα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην αγορά ήρθαν διάφορα λογότυπα, διαφορετικοί τρόποι εντοπισμού της ποιότητας, άλλα είχαν να κάνουν με τις διατροφικές ιδιότητες, άλλα είχαν να κάνουν με την υγιεινή, με τις τιμές, με τη συσκευασία κλπ. κλπ. Με αποτέλεσμα τελικά ο καταναλωτής, πιστεύουμε, και αυτό δείχνουν διάφορες αξιολογήσεις που έχουμε κάνει, δείχνουν λοιπόν ότι προκαλέσαμε έτσι σύγχυση στο καταναλωτή. Οπότε, για την πολιτική ποιότητα αυτό θέλουμε. Νομίζω ότι εδώ πέρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Θέλουμε δηλαδή εδώ να δείξουμε ποια είναι τα μέσα που έχουμε για τον έλεγχο της ποιότητας, ώστε να υπάρχει κάποια τάξη στην αγορά. Έτσι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές ξέρουν ε, τι θέλουν και τι περιμένουν από τα πράγματα που βρίσκουν στην αγορά. Προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε στην πολιτική μας αυτή ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει και ένα θέμα επικοινωνίας εδώ. Οι καταναλωτές, οι αγοραστές πρέπει να ενημερώνονται για το ποια είναι η ποιότητα των προϊόντων που αγοράζουν. Αλλά αυτό με συγκεκριμένη ενημέρωση, γιατί μόνο τότε μπορούμε να περιμένουμε πως οι καταναλωτές σωστά θα εκτιμήσουν τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και μόνο αν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες μπορούν οι παραγωγοί από την πλευρά τους να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη ζήτηση από πλευράς καταναλωτών. Έτσι λοιπόν, το πρώτο βήμα που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι πρόθεσε μια πράσινη βίβλο το 1998, ζητώντας ε, πληροφορίες από τις διάφορες πλευρές. Οι αγρότες, οι παραγωγοί, πώς θέλουν να εκφράσουν καλύτερα, να εκφράζονται καλύτερα οι απαιτήσει από τα προϊόντα τους τι χρειάζεται για την εμπορία, τι αλλαγέ χρειάζονται στα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την ε, ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων και τι θα έπρεπε να γίνει, αν θα έπρεπε να γίνει κάτι, με τα πολλά και διαφορετικά μέσα πιστοποίησης που υπάρχουν ε, και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν ε, ξεκινήσαμε μια διαβούλευση με 560 συμμετέχοντες από 31 χώρες. Είχαμε απαντήσεις από διάφορες οργανώσεις, από πολίτες, από κρατικές υπηρεσίες, από πάρα πολλές χώρες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Αργεντινή. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής δημοσιεύτηκε και συζητήθηκε σε διάσκεψη που οργάνωσε η Τσεχική Προεδρία τον Μάρτιο του 2009. Νομίζω μάλιστα ότι κάποιοι από εσά ήταν παρόντες στη διάσκεψη αυτή. Το μήνυμα το οποίο μας πέρασαν όλοι όσοι συμμετείχαν στην ε, δημόσια αυτή διαβούλευση ήταν ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τις προδιαγραφές εμπορίας πρώτα απ' όλα. Ότι για να γνωρίζουν οι καταναλωτές καλύτερα τα χαρακτηριστικά των γεωργικών ευρωπαϊκών προϊόντων χρειάζεται μια ένδειξη προέλευσης στην ετικέτα. Επίσης μας είπαν ότι το σύστημα γεωγραφικής ένδειξης χρειάζεται παρετέρω διευκρίνηση. Μας είπαν επίσης ότι το σύστημα για τα ειδικά παραδοσιακά προϊόντα πρέπει να παραμείνει και θα σας πω ποια είναι η θέση της Επιτροπής από αυτού σε λίγο και ότι πρέπει επίσης να βελτιώσουμε την λειτουργία των συστημάτων πιστοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη δικιά του την πλευρά που συμμετείχε με τη συζήτηση που η κυρία Πετρέ υπέβαλε πέρυσι. Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια συμπίπτουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ε, με το μήνυμα που πήραμε απ' έξω. Επιμένει δηλαδή στο ότι χρειάζεται ε, να αναφέρεται η προέλευση του προϊόντος, χρειάζεται επίσης ένδειξη για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση ότι επίσης χρειάζεται απλοποίηση των προδιαγραφών εμπορίας, αλλά όπου δικαιολογείται να παραμείνουν. Επίσης ότι οι διαδικασίες όσον αφορά την γεωγραφική ένδειξη χρειάζονται αναθεώρηση και προτείνεται μάλιστα και δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας γεωγραφικής ένδειξης. Όλα αυτά λοιπόν όπως σας είπα συμφωνούν με το μήνυμα που μας ήρθε απ' έξω από τον κόσμο. Το θέμα της πιστοποίησης επίσης, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να το ξαναδούμε. Με όλα αυτά λοιπόν και έχοντας συλλέξει λοιπόν τις απόψεις των κρατών μελών, των διαφόρων ε, οργανώσεων και οργανισμών του κόσμου που συμμετείχε στη διαβούλευση, με όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο που μας πέρασε ετοίμασε μία ανακοίνωση με στόχο να υπάρχει καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές, να υπάρχει απλοποίηση επίσης των διαφόρων μέσων που αξιολογούν την ποιότητα και ε, προκειμένου να βελτιωθεί οτιδήποτε έχει να κάνει με το σύστημα αξιολόγησης ώστε να έχουμε ε, προϊόντα ποιότητας. Προτείναμε επίσης κάποιους προσανατολισμούς. Αυτό για να πετύχουμε ακριβώς τους στόχους μας. Οι προσανατολισμοί αυτοί συνοψίζονται ως εξή. Πρώτον, όσον αφορά τις απαιτήσει για την παραγωγή. Οι περισσότεροι, και συμφωνεί και η Επιτροπή σε αυτό, λένε ότι δεν είναι επιθυμητή μία ετικέτα η οποία να ξεφεύγει από τις βασικές υποχρεώσεις. Θέλουμε στην ετικέτα να αναγράφεται ο χώρος παραγωγής και να τηρούνται οι προδιαγραφές εμπορίας. Αυτές όμως πρέπει να απλοποιηθούν. Ξεκινήσαμε από πέρυσι λοιπόν, ιδιαίτερα στα απορροκυπευτικά, με στόχο να έχουμε κάποιες βασικές προδιαγραφές εμπορίας σε όλους τους τομείς όπου δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε πιο πέρα, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αλλά εδώ μπορούμε επίσης να σκεφτούμε και κάποιους όρους που να χρησιμοποιούν σε θελοντική βάση φορείς. Συγχρόνως δεν πρέπει να ξεχνάμε τι δουλειά γίνεται σε διεθνές επίπεδο προς την ίδια κατεύθυνση. Γιατί οι προδιαγραφές εμπορίας είναι ένα μέσο που δεν πρέπει να εμποδίζει αλλά να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο. Γνωρίζετε ότι δουλεύουμε για το κόντεξ αλιμεντάριους, για παράδειγμα. Υπάρχει επίσης οικονομική οργάνωση των κλπ. όπου συμμετέχουμε κι εμείς. Όσον αφορά τώρα τη γεωγραφική ένδειξη, εδώ συμφωνούμε για το ότι χρειάζεται αναθεώρηση και διευκρίνηση. Κάποια σημεία προτείνουμε να αλλάξουν. Να βάλουμε δηλαδή κάποιες κατευθυντήρες γραμμές, όπως για παράδειγμα τη χρήση των πρώτων υλών στα μεταπημένα προϊόντα. Επίσης σε κάποια άλλα σημεία ίσως χρειάζεται κάποια νομοθετική πρόταση. Προς το παρόν έχουμε τρία συστήματα, τρεις κανονισμούς για τον Νίνο, τα λικέρ και τα τρόφιμα αγροτικής προέλευσης. Εδώ ίσως θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ενοποίηση, ώστε να είναι πιο απλοποιημένη η κατάσταση τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Δεν πρέπει συγχρόνως να ξεχνάμε τις συζητήσεις που γίνονται σε διεθνές επίπεδο, γιατί συζητούνται πράγματα όπως είναι η πραγματική ιδιοκτησία και πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις διμερείς συμφωνίες στις οποίες συμμετέχουμε. Αυτή την εποχή έχουμε με την Ελβετία, με την Κορέα ε, διαπραγματεύσεις για την, προστασία των γεωργικών προϊόντων. Έρχομαι τώρα στη βιολογική γεωργία. Εδώ ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε και να βελτιώσουμε βέβαια την αγορά αυτή. Εδώ η νομοθεσία είναι σχετικά πρόσφατη μόλις έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί κανονισμοί από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εφαρμοστική. Η εσωτερική αγορά είναι κατακαιρματισμένη. Ε, Ξαρτάται κατά πόσο υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση, αν υπάρχουν διαφορετικές εθνικές προδιαγραφές, αν υπάρχουν διαφορετικοί λογότυποι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως στην ανακοίνωσή της προτείνει αξιολόγηση της κατάστασης, παρακολούθηση της εξέλιξης και να έχουμε έναν ενιαίο λογότυπο ευρωπαϊκό από τον Ιούλιο του 2010 για όλα τα βιολογικά προϊόντα. Για τα παραδοσιακά προϊόντα τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό είναι ένα μέσο που προτάθηκε χωρίς να δώσει τα αποτελέσματα που επιθυμούσαμε. Έχουμε 22 τέτοια παραδοσιακά προϊόντα ε, καταγραμμένα, για το οποίο υπάρχει εγγύηση δεν υπάρχουν υποψηφιότητες πολλές, κάπου 20. Είναι ένα σύστημα περίπλοκο. Επιτρέπει την προστασία της ονομασίας ή όχι για τον εντοπισμό των παραδοσιακών προϊόντων στα κράτη-μέλη και πιστεύουμε ότι έτσι τα κράτη-μέλη όντως είναι σε καλύτερη θέση για να προστατέψουν και να προωθήσουν τα παραδοσιακά τους αυτά προϊόντα. προτείνουμε επίσης να διασφαλίσουμε τη συνοχή ανάμεσα στα όσα προτείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η fair trade κλπ. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή μεταξύ τους. Επίσης θέλουμε κατευθυντήριες γραμμές για την λειτουργία των εθνικών συστημάτων πιστοποίησης, είτε σε ιδιωτικό επίπεδο είτε σε εθνικό επίπεδο. Αυτό μας ζήτησε ο κόσμος, η διαβούλευση που κάναμε, αυτό διαπιστώσαμε, ότι λείπει διαφάνεια μερικές φορές. Υπάρχει κάποια ανισορροπία θα έλεγα. Ένα κατακλείδι. Η ανακοίνωση έχει 7 στρατηγικές γραμμές για την βελτίωση της επικοινωνίας τελικά ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και προκειμένου οι γεωργοί να μπορέσουν να βελτιώσουν ακόμα τα προϊόντα τους. Χρειάζεται συνοχή, είναι ένας όρος κλειδί στην ανακοίνωση αυτή. Για τη συνέχεια, για τα επόμενα στάδια, και ήδη μέσα στο 2009 πρέπει να κάνουμε τις αξιολογήσεις αντικτύπου για να προχωρήσουμε με τις νομοθετικές προτάσεις που θα έρθουν το 2010. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να συζητήσουμε μαζί σας ήδη υπό το νέο καθεστώς συναπόφασης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι σας τα είπα πολύ γρήγορα και πολύ συνοπτικά όσα περιλαμβάνονται στην ανακοίνωσή μας για το θέμα πολιτικής ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, μία ιδέα που είναι κάτι το τελικά έχει να κάνει η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων με τις επιθυμίες και με τις δυνατότητες των παραγωγών και των καταναλωτών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε καλή ποιότητα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό εξαρτάται και από τις προοπτικές, από το τι θέλει ο καθένας. Ίσως ποτέ να μην φτάνουμε στο ύψος των προσδοκιών. Προσπαθούμε πάντως και θέλουμε τη συνεργασία μαζί σας και με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Αυτά προς το παρόν και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ την κυρία Μπενίτε Σάλλας για αυτή την παρέμβασή της. Πρέπει να σας πω, δίνοντας το λόγο στον Τζαν Κάρλο Σκότα που θα παρουσιάσει την έκθεσή του, ότι το θέμα με το οποίο ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θέμα της ποιότητας, είναι θεμελιώδες το συζητούσαμε και το πρωί βάσει μια πρωτοβουλία του κ. Ντεντέν και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέλουμε πολύ διότι η προηγούμενη έκθεση του κυρία Πέτρε που υιοθετήθηκε στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου δεν φαίνεται να έγινε αποδεκτή και να λιευθεί και υπόψη από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ε, συνεργασία μεταξύ ημών Επιτροπής Γεωργίας ε, του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι άκρως ευαίσθητα θέματα. Το θέμα της προέλευσης. Το θέμα της προέλευσης είναι σημαντικότατο ζήτημα, διότι δεν είναι μόνο χρήσιμο για τους γεωργούς, αλλά είναι χρήσιμο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες το να γνωρίζουν αν αυτό που καταναλώνουν πραγματικά παράγεται σε συγκεκριμένη περιοχή ή αν προέρχεται από άλλες χώρες. Δεν θέλω όμως να κάνω εγώ την έκθεση, να δώσω το λόγο στον Τζαν Κάρλο Σκότα για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Έχει το λόγο Τζαν Κάρλο, ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Το θέμα των πολιτικών των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων έχει θεμελιώδη σημασία για να δοθούν οι σωστέ ε, πληροφορίες στον αγοραστή και τον καταναλωτή όσον αφορά τα χρηστικά του προϊόντος, ούτω ώστε με υπάρχει εγγύηση ότι η αγορά προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι αγοράζει κανεί προϊόντα υψηλής ποιότητας που απορρέουν από τις διάφορες περιφερειακές παραδόσεις. Θα πρέπει λοιπόν να εκπαιδευτεί ο καταναλωτής να κάνει με επίγνωση την επιλογή του. Συνεχίζοντας τις εργασίες που έκανε η Μαρία Πέτρε με την έκθεση για την ποιότητα των προϊόντων που υπευλήθη τον περασμένο Φεβρουάριο ε, θέλω και εγώ να αναλύσω κάποιε προβληματικέ που συμπεριλαμβάνω στην έκθεσή μου. Πιστεύω αναγκαίο να μπει η ετικετοθεσία προέλευση, να καταστεί υποχρεωτική στι πρώτε ύλε και να είναι κεντρικό μέσο τη πολιτική ποιότητα, διότι είναι θεμελιώδε αυτό για να εγγυηθούμε να δώσουν περισσότερες εγγυήσει στον καταναλωτή. Η ένδειξη προέλευση θα επιτρέψει ε, στον καταναλωτή ε, να έχει περισσότερες πληροφορίες και να είναι διαφανείς οι πληροφορίες και είναι απαραίτητε πληροφορίε για να κάνει επιλογέ αγορά ε, συνειδητέ. Όσον αφορά τι γεωγραφικέ ενδείξει, πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να παραμείνουν τα σχήματα ε, του καθορισμού ε, τόπου προέλευση προστατευμένου ένδειξη προέλευση και γεωγραφική, προστατευμένη ε, γεωγραφική προέλευση, ένδειξη προέλευση. Και Βεβαίωση ιδιαιτερότητε. Αντίθετα από αυτό που εξέφρασε στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων COM234, που ήθελε να συγχωνεύσει με τα μέσα DOP και AGP. Η δημιουργία ενό ενίου συστήματο προστασία θα οδηγούσε σε καλύτερο έλεγχο των προϊόντων προέλευση και θα ε, συνέδε περισσότερο το προϊόν με τη ζώνη παραγωγή. Οι κανόνε παραγωγή, μεταποίηση και κατεργασία των γεωργικών προϊόντων θα εφαρμόζονται καλύτερα. Πιστεύω ότι η πολιτική τη ποιότητα είναι θεμελιώδε στοιχείο για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών εδαφών και θα οδηγούσε σε ενίσχυση τη προστασία των αναγνωρισμένων προϊόντων μέσω της πρόβλεψης της υποχρέωσης προστασίας εξοφίσεω των ονομασιών των προστατευμένων για να εφαρμοστούν οι παρεμβάσει, πρέπει να ενισχυθούν και τα μέσα τα κατάλληλα που αξιοποιούν και ενισχύουν οικονομικά ε, όλο τον τομέα. Γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω εισαγωγή μια σαφή ένδειξη και ταυτοποίηση του δικαιούχου του δικαιώματο πνευματική ιδιοκτησίας ε, και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν κατευθυντήριε γραμμέ γραμμές για την χρήση των γεωγραφικών ενδείξεων που όπως είναι τα συστατικά επίσης πάνω στις ετικέτες του μεταποιηθέντο προϊόντος. Τέλος, για να προστευτεί το σύστημα διαχείρισης και ο αριθμός των αναγνωρισμένων ονομασιών προέλευσης προτείνω την εισαγωγή ενό επίπεδου εθνικού προστασία για να δώσει απάντηση στην άνηση παραγωγή και στι τοπικέ πωλήσει όπου ε, θα ήταν, να έχουμε ονομασίες προέλευση σε τοπικό επίπεδο θα ήταν κάτι πολύ επαχθές. Καλό τους συναδέλφους να μου κάνουν προτάσεις ούτως ώστε ε, και να με ειδοποιήσουν για τυχόν συστάσεις οι προτάσεις που έχουν εδώ και σε άλλα βήματα. Ξεκινάμε την συζήτηση. Έχουμε έξι που ζήτησαν το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Να δώσουμε το λόγο Ερνάνες Καρσία, η πρώτη αγορήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Σκότα και τους δύο για τις παρουσιάσεις τους. Σε αυτή την έκθεση εγώ βλέπω δύο πράγματα. Το ένα είναι η εσωτερική δουλειά που έχει να κάνει με την ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αν υπάρχει ονομασία προέλευση ή όχι κλπ. Και από την άλλη μεριά, πώ όλα αυτά φτάνουν στον καταναλωτή. Γιατί ο καταναλωτή έχει πρόβλημα. Και όπως είδαμε και πριν στις διαφάνειες, υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί λογότυποι που όσο υπέροχοι κι αν είναι, τελικά ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η ιδέα της απλοποίησης, της απλούστευσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ενοποίηση. Για παράδειγμα, στο σημείο που αναφέρονται οι γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασία προέλευσης, για μένα δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα γίνει αυτή η συγχώνευση συστημάτων. Μήπως θα γίνει σε βάρος της ποιότητας κάποιων προϊόντων εάν πέσουν οι προδιαγραφές ποιότητας. Γιατί βλέπετε ότι κάθε φορά που θέλουμε να απλοποιήσουμε έχουμε την τάση να ισοπεδώνουμε προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Αυτό είναι σε βάρος της εικόνας τελικά που σχηματίζει ο καταναλωτής. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Επίσης, η απλοποίηση δεν σημαίνει ενοποίηση όπως σας είπα πριν. Όταν μας μιλήσατε για διαφορετικούς τομείς όπως είναι ο ίνος, ε, τρόφιμα ή αλκοολούχα ποτά, καταλαβαίνετε ότι αν αυτοί οι τομείς ενοποιηθούν, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρχει πια διαφοροποίηση και διαφορετική μεταχείριση. Όπως είπε και ο συνάδελφος Σκότα, προσοχή. Μην ξεχνάμε τις ιδιαιτερότητες του κάθε προϊόντος. Τέλος, και αυτό νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό. Ωραία. Η αγορά, ο καταναλωτής, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, ναι. Γι' αυτό όμως και χρειάζεται να υπάρχουν διακριτικά στοιχεία, ίσως όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά πρέπει να παραμένει η διαφοροποίηση. Αυτό που χρειάζεται είναι βελτίωση του μορατού, το πώς βλέπει ο κόσμος τα προϊόντα, η προβολή των προϊόντων αυτών. Κάποιοι θέλουν μια εξωτερική υπηρεσία, έναν οργανισμό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύεται η γεωγραφική ένδεξη και η ε, ονομασία πρόλευσης. Προσοχή όμως. Κάθε φορά που φτιάχνουμε έναν οργανισμό Ξέρουμε ότι είναι πολύ επίμαχο το θέμα. Με αυτό που θα συμφωνούσα είναι ο οργανισμός που υπάρχει για την ασφάλεια τροφίμων να αναλάβει και αυτή την αρμοδιότητα με ένα νέο τμήμα ή κάποιο τμήμα της που ήδη υπάρχει και θα μπορούσε να το αναλάβει. Οπότε, ναι, να προστατευτεί περισσότερο η γεωγραφική ένδειξη και ονομασία προέλευσης. Και πάνω απ' όλα, να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή προς το καταναλωτή. Έρχομαι τώρα στο θέμα της πιστοποίησης. Η Επιτροπή λέει ότι θέλει οικολογική σήμανση για τα μεταπημένα προϊόντα ή για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, που αυτά είναι βέβαια πολύ δύσκολα ζητήματα. Όμως, εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να προσθέσουμε και την ολοκληρωμένη γεωργία, γιατί έτσι υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια για τον καταναλωτή και καταλαβαίνουμε πώς προβάλλουμε καλύτερα και περισσότερο την αξία των ευρωπαϊκών προϊόντων απέναντι στα άλλα. Καλύτερο επίσης μάρκετινγκ για τον καταναλωτή. Γι' αυτό δεν δουλεύουμε. Οπότε, η απλοποίηση των προδιαγραφών εμπορίας για το προκυπευτικά εμένα με τρομάζει κάπως. Ο κανονισμός με αυτά που λέει ελοχεύει κινδύνους. Και οι αγρότες που ασχολούνται με τον τομέα αυτόν νιώθουν ότι υπάρχουν προβλήματα με τις διαφορετικές ρυθμίσεις. Τα διάφορα καθεστώτα πρέπει να έρχονται στην... στο ίδιο επίπεδο και να ισχύουν τα ίδια για τις 27 χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλούς έχουμε γεγραμμένους για να πάρουν το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι. Λάνζ. Η κυρία Λάνζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα πράγμα θέλω να πω. Είχα τέσσερα, αλλά σε ένα θα σταθώ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να υπάρχει η εγγύηση για τις παραδοσιακές, ε, τα παραδοσιακά προϊόντα. Ναι, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Πώς θα το λύσουμε αυτό με τις προδιαγραφές της εμπορικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμένα μου φαίνεται περίεργα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι λάθος να πούμε ότι τα εθνικά, τα κράτη δηλαδή, θα προστατεύουν τα εθνικά παραδοσιακά προϊόντα και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό, γιατί με ορισμένα, για το τυρί, για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει, να υπάρχει σε ένα κράτος μόνο. Είναι πολλοί οι αγρότες που κινδυνεύουν από αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον εισηγητή να ζητήσει να προστατεύονται και αυτά τα προϊόντα όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση στο γαλακτοκομικό τομέα, λέμε να προστατεύουμε τους αγρότες μας, ναι, αλλά όχι με την πολιτική που ακολουθούμε. Γι' αυτό θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξει αυτό που αναφέρεται στην έκθεση και από τον εισηγητή θέλω να ζητήσω να εξακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προστατεύεται παραδοσιακά προϊόντα τον ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή είναι κεντρική σημασία για την γεωργία στην Ευρώπη. Με την κατάργηση των ποσοστώσεων του γάλακτος για παράδειγμα απελευθερώνεται η γεωργία, θα υπάρχουν τομείς όπου οι γεωργοί θα καλούνται να παράγουν με τιμές παγκόσμιου εμπορίου και δεν είναι δυνατόν αυτό. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος σε προϊόντα ποιότητας. Οικοδομούμε κάτι και πρέπει να οικοδομηθεί σωστά. Θα τονίσω δύο πράγματα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αυτοδεσμευτούν και οι γεωργοί με ένα διεπαγγελματικό τρόπο. Πολλά από τα προϊόντα για τα οποία συζητούμε είναι μεταποιημένα προϊόντα. Πρέπει να αποφύγουμε να συμβεί και εδώ αυτό που έγινε στο συζήτημα που συζητούσαμε πριν. Δηλαδή η προστιθέμενη αξία να παραμένει στη μεταπιατική βιομηχανία και να μην ε, απολαμβάνουν τίποτα οι γεωργοί. Οι πρώτες ύλες, η τιμή των πρώτων υλών έχει μειωθεί εν μέρη. Αυτό πρέπει να οδηγήσει ωφέλεια και των γεωργών. Αν μην μείνει το κέρδος αλλού και η πρώτη ύλη πρέπει να συνδέεται με την περιοχή στην οποία παράγεται. Αν δεν τα καταφέρουμε, αν το καταφέρουμε αυτό, εν τέλει ο Γεωργός δεν πρόκειται να υποφεληθεί. Το δεύτερο, το οποίο <clears throat> το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί σε μια συνάντηση, είναι και ο ποσοτικός έλεγχος. Γνωρίζω ότι στην Κομισιόν πολλοί δεν θέλουν να ακούσουν τέτοια πράγματα. Αλλά όταν μιλούμε για προϊόντα με χαρακτηρισμό η ονομασία προέλευσης, θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο σύστημα, κάποιος μηχανισμός ποσοτικού ελέγχου. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν πώς μπορεί να γίνει αυτό. Και βεβαίω να μην αντιβαίνει στις, ε, στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Στεφάν Λεφόλ επόμενος. Και μετά και ο Σταμπάτζη. Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρος όσον αφορά τους στόχους και συμμερίζομαι αυτά που είπε ο εισηγητής. Η Κομισιόν πάντα θέλει να πλουστεύει. Κανονικό είναι αυτό, σωστό. Αλλά σε τέτοιο θέμα υπάρχουν πολλά επίπεδα. Το επίπεδο που αφορά τη σχέση γεωργικού προϊόντος με, το, με την περιφέρεια, με την ύπεθρο. Μετά, συσχετισμός γεωργικής παραγωγής και προδιαγραφές για την παραγωγή. Και μετά όλα όσα σχετίζονται με τις προδιαγραφές, με τα πρότυπα που συνδέονται με αυτά που επιβάλλουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους γεωργούς. Τρία επίπεδα. Δεν μπορούμε, και το λέω ξεκάθαρα αυτό, δεν μπορούμε να θέλουμε να πλουστεύουμε και να θυσιάζουμε. Η γεωργία έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν έχουμε μόνο μάρκες, αλλά έχουμε και σήματα που συνδέονται με περιοχές και ποιότητα προϊόντος. Και αυτό είναι ουσιαστικό. Στην έκθεση θα ήθελα αυτό να αντικατοπτρίζεται. Εκεί να είναι προστιθέμενη αξία. Θα υποβάλω σχετικά τροπολογίες. Ηρίστον παρόδο. Η Ευρώπη έχει περισσότερους γεωργούς, λιγότερες εκτάσεις από τις ΗΠΑ και έχει μια άμυση με δύο φορές παραπάνω προστιθέμενη αξία από τις ΗΠΑ. Διερωτηθείτε. Γιατί συνδέεται με τη δυνατότητα που έχουμε να παράγουμε προστιθέμενη αξία δημιουργώντας τον κατακαιρματισμό στην αγορά. Είναι αυτή η πολιτική που πρέπει να υπερασπιστούμε, τουλάχιστον εγώ όσον αφορά αυτή την έκθεση, αυτό πρόκειται να υπερασπιστώ. Ευχαριστώ Στεφάν, ο Ταμπάτζη και μετά Δεντέ, Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι θέμα πολύ σημαντικό για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής διότι η διαφάνεια, η ενημέρωση που θα είναι μεγαλύτερη για τους καταναλωτές είναι θέμα κλειδί, ξεκάθαρα τα πράγματα. Και φοβάμαι ότι κάποιοι συνάδελφοι συγχύουν δύο πράγματα. Απ' τη μια, χρειάζεται, χρειάζονται περισσότερα κοινοτικά στοιχεία όσον αφορά το σήμα, την ετικέτα. Και παραδείγματο χάρη στη βιολογική παραγωγή υπάρχουν τόσα σήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμποδίζουν την εμπορευματοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να συγχαίουμε δύο πράγματα. Προσπάθειες για περισσότερα κοινοτικά σήματα από τη μία πλευρά, για περισσότερα κοινοτικά labels και περισσότερες γεωγραφικές ενδείξεις που είναι μια επιθυμία σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει των ανθρώπων. 60% των ανθρώπων ζητούν περισσότερες ενδείξεις προέλευση των προϊόντων. Προέλευση συγκομιδής, καταγωγή της παραγωγής των μεταπιθέντων προϊόντων, που εκεί είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Από... Προτείνω λοιπόν περισσότερα σήματα ετικετοθεσία κοινοτική και περισσότερες ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης. Για μεγαλύτερη διαφάνεια, πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για τον αγοραστή. Ποια είναι η προέλευση του προϊόντος, του τροφίμου. Εδώ δεν υπάρχουν αντιθέσεις, αντιφάσεις. Υπάρχει μια αντίθεση, αντίφαση μεταξύ απλουστεύσεως του συστήματος και περισσότερων πληροφοριών από την άλλη ορθών πληροφοριών που θα παρέχονται στον αγοραστή. Χρειάζεται εξισορρόπηση των δύο στόχων. Απλούστευση χορήγηση πληροφοριών. όπως είναι η ένδειξη γεωγραφικής προέλευσης. Ευχαριστώ κύριε Ταμπάτζη. Νταντέν και ακολουθούν οι άλλοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλά κάνατε που αναφερθήκατε στην πρωινή συνεδρίαση. Είχαμε πάνω από 100 εκπροσώπους προϊόντων που ζητούσαν ονομασία προέλευσης και γεωγραφικής προέλευσης. Απέρευσε ενδιαφέρον πόρισμα το πρωί. Απασχόληση που συνδέεται με αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή. Δείχνει η μελέτη ότι για 100.000 κιλά γάλακτος απασχολούνται 0,76 μονάδες εργαζομένων στην Τανόνε. Στα προϊόντα γαλακτοκομικά γάλακτος Αγελάδας ή τυριού έχουμε 2,1 εργαζομένους για 100.000 τόνους. 7,1 στο πρόβιο γάλα, 7,1 εργαζόμενοι για 100.000 ε, κιλά. Άρα η οικονομία ολόκληρης περιοχής ενεργοποιείται για την παραγωγή αυτή των προϊόντων. Δεν πρέπει να μειώσουμε αυτή τη διάσταση, την ποιοτική, μέσω απλής προσεγγίσεως που στρέφεται γύρω από το προϊόν, ιδιότητες που έχει όσον αφορά την υγεία. Αλλά να δούμε πώς γίνεται η παραγωγή. Πολύ συχνά τα προϊόντα με σήμα ποιοτικό παράγονται σε δύσκολες ζώνες όπου οι άνθρωποι επί σειρά ετών πολεμούσαν για να βρουν μια λύση για να μπορέσουν να μείνουν στο, στην περιοχή τους. Με την πάροδο του χρόνου απέκτησε αξία το προϊόν, απέκτησε φήμη το προϊόν. Δεν τυχαίο ότι απέκτησε φήμη ένα προϊόν είναι θέμα εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτού και παραγωγού που οδηγούν στη φήμη του προϊόντο. Αυτή η εμπιστοσύνη βέβαια πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να την εγγυόμεθα ότι υπάρχει ένα αίτιο δημιουργείται εμπιστοσύνη. Πρέπει να διονυστούν οι πολιτικές διασφάλισης ποιοτικών προϊόντων. Και για να ανοίξει, βλέπουμε ότι ανοίγει η αγορά των αγροτικών προϊόντων και φτάνουν από άλλε υπήρου προϊόντα. Εκεί πρέπει να παίξει ρόλο η ιδιαιτερότητα των προϊόντων. Να τα προστατεύσουμε. Η τεχνογνωσία που θα προστατεύσουμε είναι ένα ατού, πλεονέκτημα που οδηγεί σε προστιθέμενη αξία. Και έτσι θα παραμείνουν και οι θέσει αυτέ ε, απασχόληση που δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν από μια συγκεκριμένη περιοχή σε άλλη. Ευχαριστώ, Ντεντέ. Και μετά η κυρία Mm. Σας ευχαριστώ. Η συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας, γεωγραφικής ονομασίας κλπ. είναι σημαντική για τις τοπικές κοινωνίες και αποτελεί και μια μορφή έκφρασης για την δυναμικότητα ανάπτυξης μιας τοπικής κοινωνίας. Αυτό εξηγεί και για ποιο λόγο οι εγκρίσει κυκλοφορία τέτοιων προϊόντων καμιά φορά χρειάζονται χρόνια. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε να επιταχυνθούν διαδικασίες. Αφενός έχουμε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία είναι χαρακτηριστικά μιας τοπικής αγοράς, μπορούν να είναι και ε, ευρύτερα γνωστά τα προϊόντα αυτά. Καμιά φορά έχουν και μια ιστορική διαδρομή. Άλλο πρόβλημα είναι η προέλευση τροφίμων προϊόντων των οποίων η ακριβής προέλευση δεν είναι γνωστή. Εμείς θέλουμε βέβαια να μειώσουμε την ένταση της παραγωγής. Για παράδειγμα, ε, το γάλα να παράγεται από αγελάδες που βόσκουν σε βοσκοτόπια. Αυτό θα οδηγήσει και σε αύξηση των τιμών βέβαια, αλλά πρέπει να δοθεί η δυνατότητα αυτή στους ε, αγρότες και μάλιστα και να προαχθεί με ειδικές ενέργειες, ώστε να υπάρξει ένα νέο επίπεδο παραγωγής. Η παραγωγή των προϊόντων τροφίμων με μικρότερη για παράδειγμα χρήση λιπασμάτων ή ε, εντομοκτώνων και ζυζανιοκτώνων είναι ένας τρόπος για να αυξηθούν εν τέλει και τα έσοδα των γεωργών. Και εδώ πάντως χρειάζεται διαφάνεια. Ευχαριστώ. Πόλσον και Λάιον οι επόμενοι δύο μιλητέ. Η κυρία Πόλσον. Πρόεδρε, η έννοια της ποιότητας είναι κάτι δύσκολο. Εδώ και δέκα χρόνια ξεκινήσαμε τη δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ασφαλή τρόφιμα, ασφάλεια τροφίμων. Η έννοια της ποιότητας είναι βέβαια σημαντική. Συχνά όταν συναντώ τους εκλογείς μου, μου λέγουν θέλουμε ε, μια ετικέτα που θα αναφέρεται στην προστασία των ζώων. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στις ετικέτες που θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Παραδείγματο χάρη, κάποιοι, σαν και εμένα, ζουν στη Βόρεια Σκανδιναβία. Στα δάση. Γνωρίζουμε ότι τα γεργικά εδάφη ή μάλλον οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρές ότι καλλιεργούμε εκεί παραδοσιακά προϊόντα. Δεν μιλάμε για μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Δεν, δεν συζητάμε αυτές. Αυτές που παράγουν τρόφιμα σε μεγάλη κλίμακα, σε βιομηχανική κλίμακα. Εδώ αναφερόμαστε στις μικρές εκμεταλλεύσεις. Στους μικροκαλλιεργητές που φτιάχνουν το πρόβιο τυρί τους, το αφήνουν το τυρί τους να ζυμωθεί, να γίνουν ιδέες ζυμώσεις κλπ. Στη Βόρεια Σουηδία υπάρχει ένα ψάρι. Το streaming. Ένα είδος ρέγκας είναι το Sirstroming. Αλεσμένης ρέγκας είναι το υλικό προϊόν. Παράγεται σε ντόπιο επίπεδο, σε μικρή κλίμακα. Και πρόκειται περί προϊόντος που θα μπορούσε να έχει ετικέτα που θα λέει παραδοσιακό προϊόν. Σε διεθνές επίπεδο, σε εθνικό και τοπικό, θα πρέπει να μπορούμε να καθορίσουμε τα προϊόντα αυτά που αξίζουν ένα τέτοιο σήμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τις μικρές εκμεταλλεύσεις που παράγουν διάφορα είδη τυριών σε μικρή κλίμακα και άλλα προϊόντα σε μικρή κλίμακα. Να στατεύσουμε την τόπια παραγωγή πρέπει. Ευχαριστώ. Επόμενος. Εκτός μικροφώνου επόμενος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η ποιότητα του προϊόντος είναι σημαντική για μια μικρή χώρα όπως η Σκοτία που χρησιμοποίησε καλά τα συστήματα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης όπως ε, για παράδειγμα για το, σκοτικό, για το σκοτσέζικο βοδινό αλλά και, ε, ε κρέας αρνιού που έχουν οδηγήσει και σε αύξηση των τιμών που ευχαρίστω πλήρωσαν οι καταναλωτέ, αλλά και η οποία αύξηση των τιμών τελικά πέρασε και στου παραγωγού, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίση, έχουμε φτιάξει και συστήματα χωρίς πιστοποιητικών με καλύτερη εν τέλει πρόσβαση στην ε, λιανική αγορά και στους καταναλωτές. Ωστόσο, εγώ έχω κάποιες ανησυχίες σχετικά με την απλούστευση ή την συγχώνευση της γεωγραφικής πιστοποίησης. Να συγχωνευτούν σε ένα σύστημα δηλαδή. Αυτό δεν θα μου άρεσε καθόλου. Και θέλω να μου εγγυηθείτε ότι δεν θα χαθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας ορισμένων τοπικών τέτοιων συστημάτων. Αλλιώς δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε ό,τι αφορά τα συστήματα πιστοποίησης να προταθούν καλύτερα κατευθυντήρες γραμμές και όχι ε, αναγκαστικές ρυθμίσεις. Δεν μας χρειάζεται περισσότερη κανονιστική ρύθμιση στους ε, τομείς αυτούς. Αυτό που χρειάζεται είναι όντως κατευθυντήρες γραμμές οι οποίες να επιτρέψουν ισότιμο ανταγωνισμό παντού. Τέλος, η θέση της γεωργίας. για να εφαρμοστεί ε, το σύστημα πιστοποιήσεως σε όλα τα προϊόντα. Το ερώτημα είναι αν, ε, ξεφύγουμε από τα πρωτογενή προϊόντα για να πάμε στα μεταποιημένα, πώς γίνεται αυτό χωρίς να προσθεθεί σημαντικό κόστος, ε, έξτρα κανονιστικές ρυθμίσεις και ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση σε κόστος του συστήματος που δεν θα ωφελήσουν τους παραγωγούς ναι να αυξηθούν τα, ε, ο αριθμός των προϊόντων αλλά υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του συστήματος στα μεταποιημένα προϊόντα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη οδό. Δέχομαι ορισμένες από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά σε ό,τι αφορά τον γεωγραφικό χώρο του γεωγραφικούς χώρους παραγωγής των προϊόντων, των πιστοποιούμενων προϊόντων, θα χρειαστώ σημαντικές πρώτα εγγυήσει πριν να μπορέσω να συμφωνήσω. James Nicholson και Ζωζέ Μποβέ μετά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που διεξήχθη. Ευπρόσδεκτη. Καλό που γίνεται τώρα. Η ετικέτα προέλευσης θα επιτρέψει στον καταναλωτή να επιλέγει. Πολύ σημαντικό αυτό. Ε, εάν δεν δημιουργήσουμε ένα σύστημα, δεν λέω ομοιόμορφο, αλλά σύστημα συνεκτικό για όλη την Ευρώπη, οι υπεραγορές θα το κάνουν για μας, τα σούπερ μάρκετ. Και θα είναι εύκολο. Ενιαία προσέγγιση, διαφορετικά πρότυπα, μάλλον ανάλογα με τη βολή τους. Χώρες, προέλευση κλπ. όπως τους βολεύει και θα δημιουργηθούν προβλήματα. Πρέπει να καθορίσουμε κάποιες αρχές. Η γεωγραφική ένδειξη, όπως είπε ο προλαλής σας, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα επιστρέψουμε αρκετά στο θέμα. Αρκετές φορές στο θέμα. Έτσι θα πετύχουμε το στόχο μας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όπλο. Αν ποτέ μπει στην εργαλειοθήκη μας. Να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει άλλο ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο. Δεν θέλουμε αύξηση γραφειοκρατίας. Δεν θέλουμε να στραγγαλίσουμε ε, τον τομέα αντί να τον βοηθήσουμε. Αυτή είναι η προσέγγιση. Μπορούμε όμως να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο μόνο προσεκτικά και θα έλεγα και με κάποια ευελιξία, διότι διαβλέπω δυσκολίες σε κάποιες ε, περιοχές, σε κάποιες χώρες με... και χρειάζεται ευελιξία, ούτω ώστε όλοι να κερδίζουν. Είναι θέμα ελέγχου εισαγωγών από τρίτες χώρες, αντί πρόβλημα εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ζωσέ Μποβέ. Θέλω να παρέμβω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Είμαι, αν δεν από την πρώτη ονομασία προέλευσης που είχαμε ποτέ στην Ευρώπη. Γιατί ήταν το Ροκφόρ, το οποίο έγινε το 95. Και χάρη σε αυτή την ευρωπαϊκή δημιουργία, οι εθνικές ονομασίες προελεύσεως γίνανε κάτι άλλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια άλλη έννοια. Και τώρα έχουμε εξελίξεις με την ΟΠΕ που δεν είναι μόνο για το τελικό προϊόν, αλλά λαμβάνεται υπόψη και ε, την παραγωγή. Οπότε Βλέπετε ότι σε αυτά τα πλαίσια η Ευρώπη μας επέτρεψε πραγματικά μια ποιοτική βελτίωση της ονομασίας προελεύσεως. Τώρα αυτό επίσης που είναι σημαντικό είναι ότι υπάρχει η γη, υπάρχουν οι παραγωγοί και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στην παραγωγή. Συγχρόνως όμως όλα αυτά πρέπει να τα προστατεύσουμε. Αλλά δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με την γεωγραφική προέλευση παραγωγής. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό έχει να κάνει με ένα τελικό προϊόν και δεν λαμβάνει υπόψη τη ζώνη παραγωγής. Μπορεί να έχουμε λοιπόν ζαμπόν που ονομάζεται μπαγιόν και το οποίο μπορεί να προέρχεται από χείρους που έχουν μεγαλώσει αλλού, στη Βρετάνη ή αλλού και όχι στην Παγιόν. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε μεταξύ τους. Και όταν ερχόμαστε στη βιολογική παραγωγή, βλέπουμε ότι ο τελευταίο σχετικός κανονισμός δημιουργεί προβλήματα για το τι τελικά θα είναι πραγματικά η βιολογική προεδρία, ακριβώς γιατί σπάει τη σχέση με τη γη. Και σήμερα έχουμε λιγότερο περιοριστικούς κανόνες για την βιολογική γεωργία, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι μπορούν να αποφεληθούν και αν και δεν συμφωνώ με τον Ζωσέφ Μπορέ, το Παρμιτζάνο Ρετζάνο είναι το πιο παλιό και όχι το Ροκφόρ. Μπεντέ, και Μπεντέ, ο επόμενο αγορητή. Posso interpelar a mesa, Sr. Presidente? A primeira denominação de origem é. Κοιτάξτε, διακόπτω. Η πρώτη ονομασία προέλευση ήταν το πόρτ από το ντόρουμ, το πόρτο, το κρασί. 1700 κάτι. 1766. Την πρώτη ονομασία προέλευσης. Ευχαριστώ. Όπως βλέπετε προκαλεί και ευθυμία το θέμα. Ήδη συνέβη αυτό στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Είχαμε συζητήσει το, το θέμα και ο φίλος μας κύριος Έμπνερ που δεν είναι δυστυχώς πλέον ευρωβουλευτής Είχε πει τότε στη συζήτηση εκείνη πότε το χείριο κρέας από την Γερμανία, τη Βαβαρία γίνεται εν τέλει σπεκ, δηλαδή ένα είδος ε, ζαμβών, του Νότιου Τυρόλου. Είχε πει έχω ταξιδέψει στο Νότιο Τυρόλο αλλά ε, και έχω δει αυτό το σπεκ, ποτέ δεν έχω δει όμως χειροστάσιο το οποίο να το παράγει ε, στο Νότιο Τυρόλο εν πάση περιπτώσει, πρέπει να προσέξουμε λίγο και συμφωνώ με τον James Nicholson να μην προκαλέσουμε νέα γραφειοκρατία. Να μην δηλαδή καθιερωθούν εδώ μηχανισμοί, διαδικασίες όπου τελικώς θα καταστεί σχεδόν αδύνατο για τις ε, γεωργικές ενώσεις να ε, δημιουργήσουν πιστοποιητικά. Εγώ είμαι βαβαρός και κοντά στην, ε, στα σύνορα με την Τσεχία. Εκεί υπάρχουν πολλές ε, μικρές ε, λίμνες όπου εκτρέφονται κυπρίνοι αυτά τα ψάρια του γλυκού νερού. Έχουμε προστατεύσει την ονομασία αυτή. Είναι καλό αυτό και αυτό με ενδιαφέρει να διατηρηθεί με όσο το δυνατόν ε, μικρότερη γραφειοκρατία. για να μπορέσει έτσι και η διαφήμιση που κάνουμε προς τον καταναλωτή να είναι αξιόπιστη. Ευχαριστώ όλους για την άκουσα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ενστερνιστεί τις προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της λάβει υπόψη τη, Εδώ θα ήθελα να ζητήσω από τον Ζακάλο Σκότα κατά πόσο θα ήθελα να ολοκληρώσει με την παρέμβασή του πριν φτάσουμε στο τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης. Άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση του συναδέλφους που έκαναν προτάσεις και ελπίζω να υπάρξει και μια συμμετοχή για να φτιάξουμε το ιδεώδες κείμενο που θα ικανοποιεί τους πάντες. Σε πολλές περιπτώσεις η ετικέτα χρειάζεται και σε κάποια προϊόντα που δεν παράγουμε εμείς, διότι δεν γνωρίζουμε από πού καταφθάνουν και όμως τα τρώμε όλα, ξεκινώντας από τα μικρά στο σχολείο, στα διαλύματα, στις μεγάλες, από μεγάλους διανομής και όταν ε, ξέρουμε από πού φτάνει το προϊόν δεν θα το τρώμε. Δεν θέλω να κάνω κάποια διαφήμιση, να αναφέρω κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. Αρνητική διαφήμιση. Καλός Τζαν Κάρλο. Θα ήθελα να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξής μας, το σημείο υπαριθμών 7, παρουσίαση του θεματικού τμήματος υποστηρίζεται από θεματική διεύθυνση, από θεματικό τμήμα που εξαρτάται από τις διαθρωτικές πολιτικές συνοχής, το τμήμα συνοχής. Είναι υπεύθυνο για την ε, διερεύνηση, για να βρίσκει ειδικού για το τομέα της γεωργίας, για να εργανώνονται εργαστήρια, συνέδρια κλπ. και να υπάρχει επαρκής τεχνικό-επιστημονική υποστήριξη για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Το τμήμα, το θεματικό αυτό είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των, μελών, ε, των μελετών που ανατίθεται προς το εξωτερικό. Είναι μελέτες που δημοσιεύονται σε διάφορες γλώσσες και είναι μεγάλη σημασία για τις εργασίες μας, διότι μετά πρέπει να διεξάγονται συζητήσεις επί θεμάτων που έχουν αναλυθεί ενδελεχώς και με σοβαρότατα στοιχεία. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ το Διευθυντή της Διευθύνσεως τον κύριο Ολιβάρες Μαρτίνες θα ήθελα να του δώσω αμέσως το λόγο για να μας παρουσιάσει τη διεύθυνση αυτή για να καταλάβουμε λοιπόν πώς μπορούμε να υποφεληθούμε στις εργασίες μας, την προετοιμασία των εκθέσεων και των παρεμβάσεών μας από αυτή τη σημαντικότατη μονάδα που μας υποστηρίζει όσον αφορά τις έρευνες που διεξάγει η Επιτροπή μας. Κύριε Ολιβάρες Μαρτίνες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε να παρουσιάσουμε μια υπηρεσία ερευνών που δουλεύει και στηρίζει την Επιτροπή σας. Ξέρω ότι είμαστε στο τέλος της συνεδρίασης αυτής, αλλά παρόλα αυτά θέλω να υπογραμμίσω κάποια σημεία και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να σας εξηγήσουν τα πιο τεχνικά ζητήματα και πώς μπορείτε να αποφεληθείτε από την εσωτερική και εξωτερική πραγματογνωμοσύνη που προσφέρουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν, και δεν ξέρω αν όλοι οι νέοι βουλευτές γνωρίζουν ότι το Κοινοβούλιο αποφάσισε το 2004 να αναδιαρθρώσει τις υπηρεσίες αρρωγής προς τους ευρωβουλευτές, ώστε μέσα σε μία μονάδα να συμπεριλάβουμε και την άμεση βοήθεια ματία των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αλλά να βάλουμε εκεί μέσα και την στήριξη τη θεματική που είναι οι μονάδες έρευνας με έρευνες που κάνουν ανταποκρινόμενοι στις δικές σας αιτήσει για μελέτες, έρευνες κλπ. προκειμένου βοηθηθείτε στο έργο σας. Πραγματικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της ποιότητας του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται όλο και περισσότερο με τεχνικά ζητήματα και έτσι χρειάζεται να γνωρίζει ποια είναι, ποιες είναι οι τελευταίες γνώσεις που έχουμε στα διάφορα θέματα που εξετάζει. Για να γίνει αυτό, αποφάσισε το Κοινοβούλιο λοιπόν να συμπεριλάβει τις μονάδες έρευνας στην δομή άμεσης στήριξης προς τους ευρωβουλευτές που υπήρχε. Συγχρόνως όμως θέλησε να φτιάξει και μια δική γραμμή στον προπολογισμό για να χρηματοδοτήσει μελέτες που γίνονται έξω από το Κοινοβούλιο. Και για να στηριχτούν λοιπόν οι εσωτερικές μελέτες αλλά και να υπάρξει διοικητική στήριξη στις ε, μελέτες που ζητάμε να γίνουν εκτός Κοινοβουλίου, προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε όσο γίνεται καλύτερα οργανωτικά. Εδώ μπορώ να σας πω ότι εγώ προσωπικά ως Διευθυντής της Διορθωτικής Πολιτικής Συνοχής είμαι υπεύθυνος για το συντονισμό των εργασιών πέντε γραμματιών γραμματείων, δηλαδή πέντε κοινοβουλευτικών επιτροπών, Αλία, Γεωργία, Περιφερειακή και Αλίας. Και εγώ έχω υπό την ευθύνη μου το συντονισμό των εργασιών που κάνουν οι θεματικές υπηρεσίες για να στηρίξουν τις δικές σας κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο κλειδί. Είναι ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ε, ειδικέ ανησυχίες τις δικές σας δεν κάνουμε ακαδημαϊκές μελέτες, ούτε πρόκειται για την ικανοποίηση των, ε, της δικιάς μας διανοητικής περιέργειας. Όχι, πρόκειται για την επιθυμία μας να ανταποκριθούμε στις δικές σας ανάγκες, στις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που μας ζητάτε εσείς να κάνουμε. Δουλεύουμε δηλαδή à la carte κατά κάποιο τρόπο βάσει των όσων εσείς μας ζητάτε για να σας βοηθήσουμε στο έργο σας. Πρέπει να σας πω κάτι εντελώς ξεκάθαρα, κυρίως για να το ξέρουν οι νέοι. Μην νομίζετε ότι οι εργασίες του θεματικού τμήματος θα βοηθήσουν σε τίποτα πολιτικά. Όχι. Εσείς κάνετε την πολιτική συζήτηση, εσείς έχετε και τις πολιτικές συνέπειες, εσείς κάνετε την πολιτική και εσείς φροντίζετε να προστατεύσετε τα διάφορα συμφέροντα. Οι μελέτες που κάνουμε εμείς, τα σημειώματα που σας ετοιμάζουμε είναι μέσα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν στην πολιτική αυτή συζήτηση. Να μην υπάρχει σύγχυση εμείς και οι συνάδελφοι στη θεματική μονάδα είναι στη διάθεσή σας, αλλά για να βοηθήσουν εσάς το έργο σας. Εσείς θα αποφασίσετε ποιες είναι οι πολιτικές ανάγκες, οι θεσμικές, τι θέλετε για να στηρίξετε το έργο σας, ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες και ποιο είναι το δικό σας πολιτικό χρονοδιάγραμμα. Εμείς φροντίζουμε οι μελέτες μας να είναι ανεξάρτητες και ουδέτερες πολιτικά και να είναι τέτοιες που να δείχνουν ε, το πόσο βοηθάμε εσάς ουδέτερα. Προσπαθούμε να φροντίσουμε η ποιότητα να είναι καλή και ό,τι τελικά σας δίνουμε, ό,τι φτάνει στο γραφείο σας, να έχει γίνει πολιτικά ουδέτερα. Ως διευθυντής έχω την ευθύνη και της οικονομικής διαχείρισης, πολύ σημαντικό και αυτό. Στα πλαίσια των εξωτερικών μελετών έχουμε μια γραμμή στον προπολογισμό, υπάρχουν μέσα, αλλά υπάρχουν και περιορισμοί. Η κυρία Ολιβέρα Γκόμες, που έχω εδώ δίπλα μου και που είναι υπεύθυνη του θεματικού τμήματος και ο κύριος Μεν που είναι ο εμπειρογνώμων μας για τα θέματα γεωργίας, θα σας εξηγήσουν τις λεπτομέρειες για το πώς δουλεύει η μονάδα μας. Πάντως, εγώ έχω την ευθύνη προστασίας των συμφερόντων του σώματος. Εγώ υπογράφω τις συμβάσει. εγώ χρησιμοποιώ τα κονδύλια. Αν υπάρξει ποτέ πρόβλημα, εγώ λογοδοτώ. Ενώπιον των αρχών του λεκτικού συνεδρίου κλπ. Εσείς κάνετε την πολιτική, εμείς διασφαλίζουμε την στήριξη στην πράξη. Τέλος, και πριν δώσω το λόγο στους συναδέρφους, ο κύριος Γερακάλ που είναι υπεύθυνο στη γραμματεία, η κυρία Ολιβέρα και ο Ολιβέρα Μασότ και εγώ ίδιος, να ξέρετε ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Πάντα, όχι μόνο σήμερα, για να διασφαλίσουμε τη στήριξη που χρειάζεστε. Τέλος, Πρόεδρε, δεν ξέρετε πόσο ευτυχής είναι οι συνάδελφοι που με βλέπουν εδώ να σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί βλέπετε είναι πολύ σπάνιο οι υπάλληλοι του σώματος να έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν με την Επιτροπή για την οποία δουλεύουν. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν Πρόεδρε και συνάδελφοι εδώ θα σας δώσω πιο τεχνικές εξηγήσεις. Παρακαλώ. Παρα... Κοιτάξτε, η τεχνογνωσία που, μας, που δίνει η διεύθυνσή μας. Δεν ήμουν εγώ. Υπάρχει διαφοροποιημένη προσέγγιση. Εργασίες έρευνας. Συνεχίζει να μικροφωνίζει ο μιλητής. Θα προσπαθήσουμε ξανά και σε ελπίζουμε. Επαναλαμβάνω, τεχνογνωσία, διαφοροποιημένη έρευνα, στήριση στήριξη σε εταιρικό επίπεδο από τους υπαλλήλου του Κοινοβουλίου και εξωτερικά έγγραφα έχουμε από πανεπιστημιακούς ή συμβούλους υψηλού επίπεδου που επιλέγονται είτε μέσω διαγωνισμών ή μέσω συμβάσεων και διαπραγματευμένων διαδικασιών. Αυτή η υποστήριξη εξωτερική και εσωτερική γίνεται διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε αξιολογήσει συνεπειών όσον αφορά τον προπολογισμό και νομοθετήματα. Υπάρχουν εργαστήρια εμπειρογνωμόνων και πάνελ έχουμε εμπειρογνωμόνων για μόνιμη υποστήριξη κυρίως τα σημαντικότατα θέματα. Και συνεχής υποστήριξη παρέχεται από τα εξωτερικά μέσα. Καλύπτονται όπως είπε και ο Σοριβάρης, από τα κονδύλια για την εξωτερική στηρίξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γίνονται σεβαστοί οι κανόνες συμβασιακοί και οικονομικοί. Υπάρχουν και εσωτερικά μέσα εργαλεία, εσωτερικά σημειώματα που ετοιμάζουν οι υπάλληλοι του Ευρωκοινοβουλίου, έρευνες, κείμενα, πληροφορίες, επίκαιρες, μελέτες που δημοσίευονται αλλού, όπως τις είπα στα πανεπιστήμια. Άρθρα γνωστών περιοδικών, εφημερίδων, στατιστικά στοιχεία που μπορούμε τακτικά να σας χορηγούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κλασικού ταχυδρομείου. Και έχουμε σημαντικό το, το άλλο εργαλείο διαδεδομένων. Τα τεχνικά δελτία, δημοσιεύσεις ετήσιες που σήμερα σε έξι γλώσσες βρίσκονται επί χάρτου και ηλεκτρονικά σε όλες τις γλώσσες της κοινότητας. Αυτά τα τεχνικά δελτία επικαιροποιούνται περιοδικά. Πώς εργάζεται το τμήμα μας εργάζεται αποκλειστικά κατόπιν αιτήματος των συγκεκριμένων κοινοβουλευτικών φορέων, κοινοβουλευτικών επιτροπών και ο πρόεδρος ή συντονιστής ζητάει το κείμενο υπάρχουν μετά το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου και διευθυντή ή γενικοί διευθυντέ του Κοινοβουλίου. Είναι οι μόνοι φορεί που μπορούν να μα ζητήσουν να κάνουμε κάποια εργασία, μια μελέτη στο εσωτερικό επίπεδο. Όσον αφορά τον προπολογισμό για εξωτερικέ μελέτε. είχαμε θετική αξιολόγηση μέχρι το 2008. Το 2009 μειώθηκε ο προϋπολογισμός λόγω αλλαγή θητεία. Το 2008 περίπου 400 400.000 ευρώ έφτασε. 2009 259.000 ευρώ έφτασε το ποσό που μας διατέθη. Για φέτος 114.000 ευρώ δεσμεύτηκαν και 58.000 ευρώ απομένουν για να δαπανηθούν. Όσον αφορά τις τελευταίες έρευνες, βλέπετε ένα μικρό κατάλογο. Ήδη παρουσιάσαμε στην Επιτροπή Γεωργίας τρεις εξωτερικές μελέτες για την Αμερικανική πολιτική. Ποιες είναι οι εξελίξεις των πολυμερών διαπραγματεύσεων για τη Γεωργία και τι γίνεται με την αύξηση του, των δαπανών στον τομέα της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας. Νέες τρεις μελέτες ζητήθηκαν από την παλιά θητεία, από την παλιά Επιτροπή Γεωργίας και συντάσσονται η πρώτη αφορά το νέο μοντέλο ενιαίας πληρωμής μετά το 2013, άλλη αφορά τις συνέπειες της γύρανσης του πληθυσμού στην Ήπεθρο Τρίτον, τι γίνεται στον τομέα των πουλερικών. Διοργανώνουμε ένα εργαστήριο για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013. Στις 10 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα. Και υπάρχουν εσωτερικά σημειώματα που διανέμονται, θα νημηθούν αυτά τα σημειώματα τι επόμενε εβδομάδε όσον αφορά τις συνέπειες τη συνθήκη της Λισαβόνας και πού βρίσκεται ο προβληματισμό για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα ακολουθήσει μετά το 2013. Στόχος του τμήματό μα είναι να σα δώσει ποιοτική τεχνογνωσία, το είπαμε αυτό, που μπορεί να σα υποστηρίξει στο πολιτικό σα έργο. Τεχνογνωσία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να σα βοηθήσει να αντιμετωπίσει σημαντικέ αλλαγέ που θα σημειωθούν στην ΚΑΠ. Εισαγωγή των κριτηρίων τη Λισαβόνα, συναπόφαση που θα είναι η συνήθι νομοθετική διαδικασία στον τομέα το γεωργικό. Σημαντική στρατηγική αλλαγή αυτή. Τέλος, όλα τα έγγραφα του τμήματός μας είναι διαθέσιμα σε χαρτί ή ηλεκτρονικά. Εδώ βλέπετε τις διευθύνσεις. Υπάρχει και ε, ένα newsletter που αποστέλλεται στα μέλη και εδώ βλέπετε την ιστοσελίδα που, ιστοσελίδες που είναι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Ολιβέρα Ρούμας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πάρα πολύ σύντομα, για να ολοκληρώσουμε, θα υπογραμμίσω κάποια στοιχεία τα οποία σας παρουσιάστηκαν ήδη. Όντως, ε, η βοήθεια και στήριξη από τις μονάδες μας προσθέτει πολλά στο έργο των ε, Ευρωβουλευτών στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει εκατοντάδες έρευνες μετά από αίτημα των Επιτροπών Πολιτισμού, Γεωργίας, Αλίας, Περιφερειακής ε, και Μεταφορών. 161 σημειώματα, πολλά briefing papers, εργαστήρια και 30 μελέτες, 40 ε, σημειώματα και 4, 4 εργαστήρια μόνο για τη δικιά σας επιτροπή και βέβαια πάρα, πολλές, ε, πάρα πολλά τεχνικά δελτία που ετοιμάζουμε πάρα πολύ συχνά. Το αποτέλεσμα είναι πολύ πλούσιο. Το έχουμε επειδή ακριβώς συνεργαζόμαστε στενά με τη γραμματεία της Επιτροπής σας και συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία. Για άλλη μια φορά επιστήνω την προσοχή σας στον προϋπολογισμό για την πραγματοσύνη μέχρι τα τέλη του 2009 50.000 ευρώ. Όσον αφορά τον προπολογισμό για το 2010, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα τη ίδια τάξη μεγέθου με εκείνον που είχαμε για το 2008, δηλαδή 400.000 ευρώ. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ό,τι αιτήσει έχετε για εκθέσει να τα υποβάλει τόσο γίνεται πιο γρήγορα στου συντονιστέ σα. Όσο πιο γρήγορα εμεί πάρουμε τα αιτήματά σα, τόσο πιο ε, καλά μπορούμε να προετοιμάσουμε τα θέματα, να ξεκινήσουμε δηλαδή τις προκαταρτικές έρευνες και άρα θα είναι καλύτερο και το αποτέλεσμα της μελέτης που θα σας δώσουμε στο τέλος. Για άλλη μια φορά είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις έχετε. Θα ήθελα, μην δώσω το λόγο σε, που, αυτούς που ζήτησαν, θα ευχαριστήσω τον Διευθυντή, τον κύριο Λιβάρας Μαρτίνες, τον Αλμπέρ Μασότ και την κυρία Λιβέρα Γκόμας, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπαν. Ήξερα ήδη τη δουλειά που κάνει το τμήμα. Με τη συναπόφαση αλλάζουν τα πάντα. Και καλό και τους φίλους συντονιστές των ομάδων να το προσέξουν, διότι όλο και περισσότερο θα πρέπει οι αποφασίσεις μας να συνοδεύονται από επιστημονική τεχνική ανάλυση, αντικειμενική ανάλυση, που όλα αυτά θα μπορούν να βοηθήσουν να γίνουν οι σωστές ε, επιλογές. Ελπίζω ότι περισσότερο θα ζητάμε να δούμε ποιες είναι συνέπειες των επιλογών, ε, των προτάσεων που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει η άποψή μας, η γνώμη μας να δίνεται υποχρεωτικά πλέον. Υποχρεώμαστε τεχνικά να εμβαθύνουμε σε θέματα, οπότε η υποστήριξή σας θα είναι σημαντικότατη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την παρουσίαση. Σίγουρα ήδη αύριο στη συνεδρίαση των συντονιστών θα μιλήσουμε για αυτό το υπόλοιπο του προπολογισμού, πώς να το εφαρμόσουμε εν ώψη των μελλοντικών μας προσπαθειών. Λουίς Σκάπουλα Σάντος έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος βέβαια της συνεδρίασης αυτής. Αλλά βλέπετε δεν μπορώ παρά να κάνω ένα σχόλιο υπέρ του θεματικού τμήματος που μας στηρίζει. Εγώ ήμουνα και πριν Ευρωβουλευτής και μάλιστα για λίγο Παρ' όλα αυτά, οι επαφές που είχα με το τμήμα αυτό ήταν πάρα πολύ θετικέ. Μπορώ λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα μπορούσα να δουλέψω όπως δούλεψα αν δεν είχα τη στήριξη του θεματικού τμήματος. Γι' αυτό συγχαρητήρια σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή και για μένα, να ξέρετε, που μπορώ να πω πόσο μας έχετε βοηθήσει και να συστήσω το τμήμα σε όλους τους συναδέρφους. Γιατί η είναι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ Λουίς, άλλος ένας. Κριστίν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική εργασία σας και έχω μια τεχνική ερώτηση. η μη εγγεγραμμένη αποκλείονται ε, γενικά από μια σειρά δραστηριοτήτων εδώ εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, εφόσον είναι ε, μια ομάδα μεταξύ των εγγεγραμμένων, ποια δυνατότητα έχουν να ε, κάνουν χρήση των υπηρεσιών σας. για παράδειγμα για να ασκηθεί ε, κάποια ε, πίεση ε, απέναντι σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν μιλάω για τίποτα το τρομερά ριζοσπαστικό, αλλά τέλο πάντων για να προστατευθούν οι ε, γεωργοί. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, όταν μείνει και γραμμένοι, θα θέλαμε να μάθουμε αυτό το πράγμα. Να, να εγγραφείτε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση από πλευρά του, της Ορίστε, είναι απλούστατο. Όπως υπόθηκε, αρκεί να απευθυνθείτε στο συντονιστή. Να στείλετε στη γραμματεία της Επιτροπής γραπτό στο έτοιμά σας, θα υποβληθεί στη συνεδρία των συντονιστών και οι συντονιστές θα αποφασίσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε πραγματικά εκ βάθους καρδίας το θεματικό τμήμα. Ευχαριστούμε όλους τους βουλευτές. Αύριο το πρωί σας θυμίζω 9 συνεδρίαση των συντονιστών, 10